Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, just, uh, Καλησπέρα σα, κύριε και κύριοι. Ε, να σα ανακοινώσω ότι ο πρόεδρο Λόπε δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Μου ζητήθηκε λοιπόν να τον αντικαταστήσω, δεν το κάνω αυθαίρετα. Mm. Είχαμε και πολύ ωραία αποτελέσματα στο Wimbledon χθε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώ ορίσατε όλοι στην απογευματινή μα συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι όσοι είστε εδώ ως εκπρόσωποι διαφορών υπηρεσιών, να είστε εδώ στις 5 το απόγευμα. Τότε ψηφίζουμε. Ενημερώστε παρακαλώ όσους συναδέλφους χρειάζεται. Καταρχάς, το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης έχει δύο μικρές αλλαγές. Η πρώτη είναι το σημείο 17 η έκθεση της κυρίας Βίξτρομ για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδέ, ανταλλαγές μαθητών, την έμιστη ή άμυστη κατάρτιση, εθελοντική εργασία και απασχόληση ως εσωτερική άμυστη βοηθή. Αυτό θα συζητηθεί αύριο στις 9 το πρωί. Αντί για τις 11. Στις 9 λοιπόν και το σημείο 11 η έκθεση του κυρίου Μισελ για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 θα συζητηθεί στις 11 το πρωί αντί για τις 9. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 2. Θα Ήθελα να σας αναφέρω τις συστάσεις των συντονιστών προς έγκριση, καταρχάς ορισμός ε, εισηγητών. Ο κύριος από το ΕΛΚ ορίστηκε εισηγητής για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την διαχείριση, συνεργασία με τρίτες χώρες και πρακτική εφαρμογή της ε, οδηγίας επιστροφής. Η κυρία Κίνγκα Γκόντς ορίστηκε η συγγήτρια για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τον πίνακα πηδώσεων της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και η κυρία Λούνα Τσέκα από τους Πρασίνους ορίστηκε η συγγήτρια για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του δικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της ομοφοβίας και των διακρίσεων βασισμένων ε, στις σεξουαλικές προτιμήσεις. Ο κύριος Νομέλο του ΕΛΚ η εισηγητή για την έκθεση Δία πρωτοβουλία με θέμα την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. και Τη ε, Αρμόδιας επιτροπή ΑΦΚΟΗ. Κατά την ε, συνεδρίαση Τη 27η Ιουνίου οι συντονιστέ αποφάσισαν να καταθέσουν δύο προφορικέ ερωτήσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εκ μέρου τη Επιτροπή ΕΛΥΜΠΕ για να συζητηθούν στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Ή το ψήφισμα για την ε, συμφωνία TTIP του Σεπτεμβρίου ζήτησε ακόλουθου ελέγχου την επόμενη χρονιά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτές τις συστάσεις των συντονιστών, μπορούμε να τις εγκρίνουμε. Εγκρίνονται λοιπόν. Περνάμε τώρα στο σημείο 3. για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετήσια έκθεση του 2012 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οργανισμός ενέκρινε την ετήσια έκθεση του για το 2012 και σήμερα υποβάλλει την έκθεση στην Επιτροπή μας όπως προβλέπεται από το άρθρο 24.6β για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με χαρά μας σήμερα καλωσορίζουμε την κυρία Σάξιν, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κύριο Κέρουμ, διευθυντή του οργανισμού. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Σάξιν και μετά στον κύριο Κέρουμ για να μας παρουσιάσουν την ετήσια έκθεση και μετά από την παρουσίαση αυτή καλούνται τα μέλη που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις να το πράξουν. Κυρία Σάξιν, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Διακεκριμένα Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αγαπητοί συνάδελφοι. Μεγάλη χαρά για μας που ήρθαμε εδώ να σας παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεσή μας. Είναι μία από τις ε, σημαντικότερες εκθέσεις ε, προϊόν του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στον ιδιωτικό κανονισμό, στο προήμιο, αναφέρει το εξής. Αναφέρει πίσω οι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδει ελευθερίε και το κράτο δικαίου και αυτές οι αξίες γίνονται σεβαστές από τα κράτη-μέλη. Η Ένωση και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλες τις δράσεις τους. Υπήρχε ανάγκη και υπάρχει ανάγκη για περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο Λενισμός. Και ένα από τα βασικά καθήκοντα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, καθήκοντά μας, είναι κάθε χρόνο να υποβάλουμε έκθεση στο Κοινοβούλιο, τον ημερώνουμε. Σημαντικότατα αυτό από την πλευρά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει το καθήκον αυτό πολύ στα σοβαρά και έχουμε εκλέξει μια επιτροπή εκδοτική που συντάσσει την αλόγο έκθεση. Και θεωρούμε σημαντικότατο το ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συζητήσει τις δραστηριότητές μας και τα επιτεύγματά μας, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συζητήσει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Στην έκθεσή μας σας παρέχουμε μία επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και βλέπετε πώς εφαρμόζεται και ερμηνεύεται αυτή στα κράτη-μέλη και αυτό είναι σημαντικότατο από την σκοπιά της δημοκρατίας, δηλαδή το Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα με τις διάφορες νομοθεσίες. Στην παρουσίασή μας θα δώσω το λόγο στον Μόρτεν Κιέρουμ, ο οποίος θα αναφερθεί λεπτομερέστερα στα διάφορα κεφάλαια. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι συμφωνείτε μαζί μας όσον αφορά τη σύσταση της επιστημονικής μας επιτροπής που η Επιστημονική Επιτροπή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο εγγυάται την υψηλή ποιότητα της έκθεσής μας, η Επιτροπή αυτή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε επίσης για την καλή συνεργασία, για την παράταση της θητείας του κυρίου Μόρτεν Κέρουμ. Προσωπικά θα έλεγα ότι αυτό είναι σημαντικότατο για μένα, όπως βλέπετε. Σήμερα βλέπετε παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω αυτή την συνέχεια της άριστης συνεργασίας μας στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ όλους σας επίσης, όλους όσους συμμετείχατε στην εξωτερική αξιολόγηση, στις συνεντεύξεις. Σημαντικότατο εγχείρημα. Ευχαριστώ που μας δώσατε χρόνο, μας αφιερώσατε χρόνο απαντώντας τις απαντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συζήτησε τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολογήσεως και συμφωνήσαμε επί προτάσεων για το μέλλον. Αποφασίσαμε πράγματα που σχετίζονται με, τα... με τον καταστατικό μας κανονισμό. Έχουμε κάποιες συστάσεις για ενδεχόμενες αλλαγές όσον αφορά τον καταστατικό αυτό κανονισμό και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις βάσει της αξιολογήσεως. Πρόθεσή μας είναι να υιοθετήσουμε νέα στρατηγική το Δεκέμβριο. Και στο μέλλον επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ιδέες μας. Τώρα όμως επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Μόρτεν Κίρμ που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που επέστρεψα εδώ να συζητήσουμε εκ νέου την ετήσια έκθεσή μας. Συνεχίζοντας και εγώ τις ευχαριστίες, ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την επίσκεψη στην Βιέννη το Φεβρουάριο. Εκτιμήσαμε πολύ αυτή την επίσκεψη, θεωρήσαμε ότι υπήρξε άριστη ανταλλαγή απόψεων. Και είχαμε και κάποιες ιδέες για ενίσχυση μελλοντική της συνεργασίας. Και τα όσα είπε και η Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την στήριξή σας, για την παράταση του, της συμβάσεώς μου. Όπως και πέρσι και φέτος, έχουμε συγκεκριμένα κεφάλαια στην έκθεση. Πέρσι εξετάσαμε τα θεμελιώδη, το τοπίο των θεμελιώδων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Φέτος υπογραμμίζουμε το πώς η κρίση επηρεάζει τον τομέα αυτό και πώς αλλάζει το τοπίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι σαφές τη σπάση ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε όμως και πολιτική κρίση. Θα το δούμε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αυτό. Και κάποιο είδους συνταγματική κρίση. Βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν διάφορες πτυχές τις ιδρυτικής συνθήκες. Το άρθρο 2, πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 6 και βέβαια οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ακροθυγός θα αναφερθώ στις τρεις διαστάσεις. Το ευάλωτο των θεμελιών δικαιωμάτων και οι παραβιάσεις των θεμελιών δικαιωμάτων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, οικονομικής κρίσης. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να βρει την άμεση σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσεως και συγκεκριμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Τα δικαιώματα των παιδιών πρώτα απ' όλα. Βλέποντας πόσα παιδιά ζουν σε, ακραία, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη και τη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, την ανεργία πλήρη της οικογένειας και τις περικοπές των προϋπολογισμών όσον αφορά τις εθνικές κοινωνικέ δαπάνες και ταυτόχρονα βλέπουμε προβλήματα για την πρόσβαση στην παιδεία, πρόσβαση στην υγεία για κάποιες ευάλωτες ομάδες, τα ευάλωτα παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση. Και άτομα με αναπηρίες. Και εκεί βγαίνουν ε, ε, εκτός των θεσμών αυτά τα άτομα. Όταν φεύγουν από κάποια ιδρύματα αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στην κοινωνία, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Χρειάζονται τοπική υποστήριξη. Και αυτή μειώνεται λόγω περικοπών. Και έτσι οι άνθρωποι ε, κινδυνεύουν, είναι πολύ ευάλωτοι και κινδυνεύουν γιατί δεν καλύπτονται. Υπάρχει και κάποια πρόοδος βέβαια στον τομέα της κοινωνικο-οικονομικής κρίσεως. Τα θύματα κυρίως. Η οδηγία για τα θύματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει προωθήσει αυτό το θέμα. Και στα κράτη-μέλη υπάρχει μια αναδιοργάνωση όσον αφορά τη στήριξη των θυμάτων. Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που παρέχεται στα θύματα. Άρα είναι ανάμεικτη εικόνα. Αλλά υπάρχουν λόγοι για ανησυχίες όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική κρίση και τη σχετική διάσταση. Να στραφώ τώρα στην πολιτική κρίση. Έχουμε διάφορες καταστάσεις που είδαμε το 2012, κρισίμου σημασίας για τα πολιτικά συστήματα. Κάποια κράτη-μέλη διαπίστωσαν κοινωνική αναταραχή, δημόσια διαμαρτυρία και κάτι που μας ανησυχεί πολύ, πρωτοβουλίες κατά των μεταναστών και μείωση της εμπιστοσύνης όσον αφορά τις εθνικές κυβερνήσεις και προς κάποιους θεσμούς εθνικούς. Κάποιες έρευνες έδειξαν έλλειψη εμπιστοσύνη στο γενικό σύστημα το δικαστικό. Τα στοιχεία τα ξέρετε που συνέλεξε ο οργανισμός μας. Οργανισμοί και ομάδες και κυρίως οι Ρωμά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω διακρίσεων και αντιμετωπίζουν και προβλήματα από βιοπραγίες. Και ανησυχούμε κυρίως διότι βλέπουμε ότι έχουμε εγκλήματα που έχουν κίνητα την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Και αυτά συμβαίνουν και στα 27 κράτη-μέλη. Ε, δύσκολο να αξιολογήσει κανείς με απόλυτους όρους το επίπεδο, αλλά οι υπολογισμοί μας μας λένε ότι δεν μειώνονται τα ποσοστά αυτών των πράξεων και πιθανότατα αυξάνονται. Αυτό είναι το πλαίσιο και έτσι εντοπίσαμε εξελίξεις που σχετίζονται με το φαινόμενο της μυσαλλοδοξίας, του εγκλήματος μυσαλλοδοξίας. Είναι βασικό θέμα, το έγκλημα μίσους, αυτό εξετάσαμε περισσότερο. Η ετήσια έκθεση βλέπει ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την διαθεσιμότητα επισήμων στοιχείων. Πώς συλλέγονται τα στοιχεία στα κάτι μέλη όσον αφορά τα εγκλήματα λόγω μίσους. Από τη διαφάνεια βλέπετε ότι μόνο σε τέσσερις χώρες βλέπουμε να υπάρχει μια πλήρης συλλογή στοιχείων. Στις υπόλοιπες χώρες βλέπουμε να υπάρχουν καλά στοιχεία αλλά οι περισσότερες χώρες δεν έχουν αρκετά στοιχεία. Πολλά πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να αυξηθεί αυτή η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θεσμικά όργανα την αστυνομία, όλους τους φορείς που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να μπορέσουμε και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αξιολογήσουμε ε, ποιες είναι οι γενικότερες τάσεις. Τελευταία διάσταση της κρίσεως που περιγράφουμε και πώς επηρεάζει τα όλα θέματα. Η συνταγματική κρίση λοιπόν αφορά το άρθρο 2 που αναφέρεται στις προκλήσεις στην έκθεσή μας. Δεξάγεται μια συζήτηση, όπως ξέρετε, σε επίπεδο κρατών μελών Προσπαθούμε να δούμε πώς οι προκλήσεις του άρθρου 2, οι συνταγματικές προκλήσεις μπορούν να αξιολογηθούν πιο εστιασμένα. Πρόσφατα θα είδατε μια έκθεση που υπευλήθη στην Επιτροπή, την έκθεση του κυρίου Ταβάρες, που τη σημειώσαμε δεόντως. Στην υπηρεσία θεωρούμε, στον οργανισμό θεωρούμε, ότι υπάρχουν πληροφορίες και θα πρέπει να συλλέγονται με πιο εστιασμένο τρόπο ούτως ώστε να λαμβάνονται πιο καλά υπόψη τα στοιχεία στις συζητήσεις. Υπάρχει περιθώριο για ε, ε, δημιουργικό πραγματισμό σε αυτό το τομέα και ο οργανισμός μας είναι έτοιμος να παίξει το ρόλο του. Μία συζήτηση που διεξάγεται εδώ είναι η εξής. Πώς η έκθεσή μας τα επόμενα χρόνια μπορεί να παίξει ρόλο στις συζητήσεις. Πώς η έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση, για την εφαρμογή του κάτους δικαίου. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω, θέλω να αναφερθώ σε κάποια άλλα στοιχεία, σε κάποιες άλλες συνιστώσεις της ετησίας εκθέσεως. Πρώτα απ' όλα, άσυλο και μετανάστευση. Ο τομέας αυτός. Το 2012 Είδαμε κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πακέτο ασύλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που υιοθετήθηκε φέτος. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να βλέπουμε έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Ένα στοιχείο να σας δώσω που αναφέρεται στην έκθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεκατέστησαν περισσότερους μετανάστες πρόσφυγες από τη Μάλτα από ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Βλέποντας επίσης και την κράτηση των ετούντων άσυλο, υπάρχει δυνατότητα εναλλακτική λύσεως από την κράτηση, που δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ, βλέποντας τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη. Τέλος, σχετικά με αυτό, για την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, περίπου το 1 τρίτο των ετούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παιδιά. Και εδώ έχουμε άλλη μια ομάδα ευάλωτων παιδιών που σίγουρα θα πρέπει να προσεχθεί και θα πρέπει να κάνουμε τα δέοντα μέσω νομοθεσίας και πρακτικής που ακολουθούμε για τη βελτίωση. Εντάχει, προχωρώ πάνω στον τομέα της ισότητας, της νομοθεσίας περισσότητας. Βλέπουμε λοιπόν το 2012 πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που επικύρωσαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και έτσι έχουμε συνολικά 25 κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την προστασία ατόμων με αναπηρίες στο μέλλον. Και βέβαια γίνεται σειρά βημάτων και στον οργανισμό και αλλού για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω συμβάσεως. Άλλη τάση όσον αφορά την ισότητα, κάτι που παρατηρήσαν το 2012. Τα κράτη έχουν θεσπίσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα νομικά καθεστώτα για την αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Βλέπουμε φορείς ισότητας όλο και περισσότερο να καλύπτουν το ζήτημα αυτό. Και τέλος, η ηλικιακή διάκριση βλέπουμε φορείς ισότητας, εθνικά δικαστήρια, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να εκδικάζουν υποθέσεις διάκρισης με βάση την ηλικία. Πιθανότατα αυτό είναι προϊόν της κρίσεως. Δηλαδή τα ηλικιωμένα άτομα απολύονται πριν από τους άλλους. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εδώ δεν βλέπουμε πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε συνδυάσει 486 αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στασβούργου που θεώρησε το δικαστήριο ότι παραβίασαν τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση το 2012. Μισές από τις υποθέσεις αναφέρονται στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη είτε δικαίωμα αποζημίωσης, δικαίωμα πρόσβασης στην δικαιοδοσία ή στο δικαίωμα δίκαιης δίκης. Άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων και σε επίπεδο 100 μελών έχουν αναλυθεί διάφορες ε, δραστηριότητες. Τέλος, η έκθεση φέτος εξετάζει το πώς συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη στις διεθνείς τους υποχρεώσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ έχουμε ομαδοποίησει τα στοιχεία που αφορούν συμβάσεις και πρωτόκολλα που έχουν γίνει αποδεκτά και βλέπουμε το χάρτη, το σχετικό. Πάντα είναι ενδιαφέρον να μην εξετάσει κανείς στατικές φωτογραφίες αλλά, της καταστάσεως αλλά και τάσεις. Να αναφέρω μια τάση που βλέπουμε. Άλλες 18 κυρώσεις από κράτη-μέλη βασικών εγγράφων του Συμβουλίου της Ευρώπης και 14 νέες κυρώσεις συμβάσεων του ΟΗΕ και πρωτοκόλων του ΟΗΕ. Τέλος, καλά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Βλέπουμε ότι πρόσφατη, πρόσφατη σύμβαση για την παραβίαση της Κωνσταντινούπολης για την παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών εκεί οι δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Ελπίζουμε η, η, έκθεση που θα κάνουμε, ετοιμάσουμε τέλος αυτού του χρόνου και αρχές του επόμενου έτους για τη βία κατά των γυναικών θα βοηθήσει να προωθηθεί η επικύρωση αυτής της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης. Εν συντομία, έδωσα μια, κάποιες εικόνες, φωτογραφίες αν θέλετε, της πληρέστατης αυτής ετήσιας εκθέσεως που ελπίζω να τη βρείτε χρήσιμη και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα κεφάλαια στην καθημερινή σας δουλειά που αφορούν τους διάφορους τομείς, τα διάφορα χαρτοφυλάκια έτσι ετοιμάστηκαν και συντάχθηκαν, όχι για να διαβάσετε την έκθεση από το α μέχρι το ω, να διαβάσετε το κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά, σαν κάτι αυτόνομο. Του χρόνου Δεν θέλω να κάνω εισαγωγή στην έκθεση του επόμενου έτους, αλλά ήθελα να πω ότι ένα από τα θέματα που θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε κεφάλαιο είναι η συνέχιση τη συζητήσεως για το κάτω δικαίου. Προχωρά γρήγορα να δούμε πού βρισκόμαστε για το συγκεκριμένο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος θέλει να συνεισφέρει επί του θέματος. Το επόμενο θέμα αφορά την αντιπροσωπεία ε, στη Βιέννη το Φεβρουάριο στην οποία αναφερθήκατε και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Γκρέιμ, ο Σερ Γκρέιμ Βότσον είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω, επειδή προείδρευσα τότε, είχα αυτή την τιμή όταν ε, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Βιέννη, ότι χαίρομαι που βρίσκεται εδώ ενώπιον μας η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διευθυντής που μας παρουσιάζουν την ετήσια έκθεση και μας δίνουν τη δυνατότητα να θίξουμε επιμέρους ζητήματα. Ο Λουί Μισελ εκφράζει την λύπη του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ο κύριος ε, Μίτσουλ δεν μπορεί να βρίσκεται, να βρεθεί εδώ μαζί μας και έχει υψηλές προσδοκίες ε, μέσα στα πλαίσια της δράσης των φιλελευθέρων για τον οργανισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αφιστεί των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως το άρθρο 7 εκεί που χρειάζεται. Και θα θέλαμε η Επιτροπή και το Συμβούλιο να είναι πιο δραστηροί στην προώθηση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ξέρω, κύριε Κέρον, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ο οργανισμός σας και να ενισχυθεί η εντολή του. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, στα πλαίσια μιας συζήτησης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συντάσει ο οργανισμός ετήσιες εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 2 στα, στην Ένωση και τα κράτη-μέλη οριζοντίως γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση που τονίζεται στη σελίδα 5 της έκθεσής σας για το 12, όταν μιλάτε για ανησυχίες για το κράτος δικαίου, ιδιαίτερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε ορισμένα κράτη-μέλη, με βάση δηλαδή το δικαστικό τομέα όπως έχει εξελιχθεί το 12, όπου αμφισβητεί τούνται ορισμένα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Αυτό έχει, αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2013 και θα θέλαμε να είσαστε πιο δραστήριοι για να υποστηριχθεί η εργασία σας σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο δεν ε, εντάσσεται στην έκθεσή σας, αλλά έχουν τεθεί θέματα αρχής. Οι διακρίσεις δηλαδή κατά των ε, Ρώσων, γιατί υπό την Προεδρία της Λιθουανίας, νομίζω η Λιθουανία θέτει το καλύτερο παράδειγμα των βαλτικών χωρών όταν μιλάει για ε, μειονότητες εθνοτήτων ως προς την εθνότητα δηλαδή των Ρώσων. Δεν ξέρω κατά πόσο ο οργανισμός σας έχει συλλέξει στοιχεία σε σχέση με την μειονότητα των Ρώσων στα βαλτικά κράτη και κατά πόσο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τη Λιθουανική Προεδρία κατά το εξάμεινο αυτό έτσι ώστε να προωθήσετε αυτό που ζήτησα και από την Προεδρεύουσα, δηλαδή τα βαλτικά κράτη να ασχοληθούν με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ε, μειονότητα, η εθνότητα των Ρώσων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Μπορούμε να δούμε όλες τις ερωτήσεις ε, και μετά εσείς να συνοψίσετε. Εντάξει. Ο κύριος Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εισήγηση αυτή τρεις-τέσσερις μήνες πριν το Φεβρουάριο συναντηθήκαμε στη Βιέννη, στην έδρα σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία σας και για τις συζητήσεις, τις ανταλλαγές απόψεων Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι παρόντες που είχαν παρευρεθεί στη Βιέννη, στην αντιπροσωπεία. Ήταν πολύ επικοδομητικό για μας, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσουμε τον οργανισμό σας για την περαιτέρω εργασία και νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας βοηθήσει στο μέλλον για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε μία ουσιαστική συνεργασία. Παρακολούθησα την ε, εισαγωγή σας, θυμάμαι και τις συζητήσεις που είχαμε τότε και η ερώτησή μου έχει ως εξής. Θυμάμαι το συζητήσαμε στη Βιέννη, έχουμε αυτό το βασικό κείμενο, αναφερθήκαμε στα κράτη-μέλη, στην εξέλιξη της κατάστασης και τις ε, βελτιώσεις σε συγκεκριμένους τομείς Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεσή σας, είναι στοιχεία ζωτική σημασίας πράγματι για την εργασία μας. Θα θέλαμε όμως και πάντα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να υπάρχει αυτός ο συσχετισμός με τα σχόλια αυτά και αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό είναι κάτι που μπορείτε να βελτιώσετε. Μπορείτε δηλαδή μέσα στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών να προωθήσετε κάτι τέτοιο. δηλαδή προτάσεις που θα μπορούσαν να προέλθουν από εσάς επί του θέματος. Δεύτερον, αυτή η διάδραση που ε, υπάρχει μεταξύ των δικών σας ε, ερευνών και σχολείων και άλλων που λαμβάνουμε από καιρού εις καιρών, δηλαδή ένα μήνα πριν, μας παρουσιάστηκε μια έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο από τα Ηνωμένα Έθνη, από τον ειδικό εισηγητή, σε σχέση με τα δικαιώματα και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ευρώπη. Και είχαν ε, συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις, στοχοθέτηση δηλαδή για την Ελλάδα και Ιταλία. Και θυμάμαι ότι ένα χρόνο πριν και εσείς συντάξατε, διενεργήσατε μία έρευνα για την Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η διάδραση μεταξύ συγκεκριμένων τομέων και εκθέσεων Δηλαδή μπορεί κάτι να είναι προσθέμενη, να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό σας, αν υπάρχει καλύτερος ε, συντονισμός. Δηλαδή ο ειδικό εισηγητής σας ενημέρωσε για την έρευνα αυτή. Προσπαθήσατε εσείς ε, επίσης να σχολιάσετε η εργασία σας μπορεί να σταθεί χρήσιμη για όλους που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα και για επιμέρους ζητήματα. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία σας στη Βιέννη, για την εργασία σας, και να είστε σίγουροι ότι από πλευράς Κοινοβουλίου και εμείς καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποδοτικά την εργασία σας και τα στοιχεία που μας ε, χορηγείτε κάθε χρόνο και όπου χρειαστεί και επιμέρους βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα άλλο μέλος της αντιπροσωπείας, η κυρία Τανόκα, θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Κέρον και την ομάδα του για άλλη μία φορά και εγώ συμμετείχα στην αντιπροσωπεία το Φεβρουάριο και ήταν άκρος ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση και η επίσκεψη και όταν κάποιος δεν ξέρει εις βάθος τα ζητήματα δεν ξέρει πώς λειτουργεί όλους ε, μηχανισμός. Εγώ βρίσκω ότι λειτουργεί πολύ καλά. Οι βασικοί περιορισμοί ενυπάρχουν στο νόμο, ο οποίος ε, ρυθμίζει αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε το πεδίο των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και εγώ είχα αναλάβει μία έκθεση ως προς συμφωνίες με το Συμβούλιο και το, ότι δεν διευρύνθηκε η εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Διαβάζοντας ε, αυτό το δελτίο, στις σελίδες 33-34 ε, για το ρατσισμό και τις εθνικές διακρίσεις γράφεται εδώ ότι δεν υπάρχουν ε, επαρκή στοιχεία από πλευράς κρατών μελών για τα εγκλήματα, ρατσιστικά εγκλήματα, ισλαμοφοβικά, κατά τον Ρωμά και ούτω καθεξής. Εμείς ως μέλη του Κοινοβουλίου και εγώ συγκεκριμένα υπέβαλα μία ερώτηση προφορική ερώτηση με ψήφισμα για τα εξτρεμιστικά εγκλήματα. και τους λόγους ε, μίσους Πώς μπορείτε να συλλέξετε αυτά τα στοιχεία. Εδώ λαμβάνω υπόψη την ε, Λετωνία και από όσο ξέρω έχουν καταγραφεί ορισμένα εγκλήματα τα οποία δεν αναφέρονται εδώ στην έκθεσή σας στον πίνακα 3. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πώς θα εντάσσετε όλα αυτά. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπρόν. Ευχαριστώ πολύ. Το πιο σημαντικό και πιο θεμελιώδες από όλα τα δικαιώματα είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Χωρίς αυτά δεν ε, γίνεται να πραγματοποιηθεί πολιτική αλλαγή και η δημοκρατία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Η ελευθερία του λόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό δικαίωμα, διότι χωρίς την ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον χωρί, ε, ανταλλαγή απόψεων που <clears throat> να είναι δίκαιη. Η αιτία, αιτήσια έκθεση Νομίζω πως δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Γιατί. Ίσως γιατί ο οργανισμός και πολλά μέλη του οργανισμού δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος ότι ο οργανισμός επιθυμεί το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου για όσους ε, συμφωνούν με αυτό. Όμως, η ελευθερία του λόγου για όσους ε, ασκούν κριτική είναι κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Και εκεί υπάρχει δαιμονοποίηση, αποκαλείται ρητορική μίσους και αναρωτιέμαι γιατί. Αυτή η έκθεση στο πίσω μέρος αναφέρεται σε αυτά τα σύνολα. Κύριε Ματσόλα, ευχαριστώ πολύ. Είμαι σχετικά νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούσα λοιπόν να είμαι μέλος της αντιπροσωπείας όταν ε, επισκεφθήκαμε τον οργανισμό στην ε, Βιέννη. Είμαι από τη Μάλτα και μου έκανε έκπληξη το γεγονός τη ε, της έλλειψης αλληλεγγύης προς τη χώρα μου ως προς τον καταμερισμό της ευθύνης. Θα ήθελα μετά από τον συνάδελφο κύριο Παπα-Νικολάου να πω και εγώ ότι η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η Μάλτα είναι μόνη της ε, όσον αφορά την, ε, το φορτίο της ε, διαχείρισης μετανάστευσης και ασύλου. Και στη σελίδα 151 στο σημείο 2 της έκθεσής σας φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. φέρετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δείξει πολύ μεγαλύτερη προθυμία να βοηθήσουν τη Μάλτα σε αυτό το θέμα. Και ως πολιτικός μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσω αυτό στους ψηφοφόρους μου στη Μάλκα. Μάλτα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στην εξή ερώτηση. Τι κάνει ο οργανισμός ή τι προτίθεται να κάνει όσον αφορά τις ε, περαιτέρω προτάσεις έτσι ώστε να βοηθήσει τη χώρα μου, να δείξει αλληλεγγύη. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οπισθοχωρήσει ως προς την προηγούμενη δέσμευσή της ε, για την ε, ε τους υποδοχής και ξέρω ότι υπήρχε αντίσταση από το Συμβούλιο, ωστόσο εσείς ως οργανισμός μπορείτε να είστε πρωτοπόροι στο να δείξετε αλληλεγγύη σε χώρες όπως η Μάλτα, έτσι ώστε να, μπορείτε να, να μπορούμε και εμείς να δικαιολογήσουμε στους ψηφοφόρους μας ότι πραγματικά κάνουμε ε, κάτι που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλάις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω μία ερώτηση όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ουδετερότητα, την πολιτική ουδετερότητα που πρέπει να υπάρχει σε αυτήν την έκθεση. Εγώ βλέπω μία αναφορά στο Front National στη Γαλλία, στην έκθεση, όπου αναφέρεται ότι το Front National είναι ένα κόμμα ξενοφοβικό κατά των μουσουλμάνων, κατά της μετανάστευσης, παρομοίως με το κόμμα της ελευθερίας στην Ολλανδία. Αυτά όμως τα κόμματα είναι και τα δύο δημοκρατικά και τα έχουν ψηφίσει πολλοί πολίτες διότι ασχολούνται με πραγματικά προγράμματα της κοινωνίας, με προβλήματα τα οποία ε, δεν ασχολούνται τα παραδοσιακά κόμματα, με τα οποία δεν ασχολείται η κυβέρνηση. Και πώς να το πω. Παρατηρώ ότι πάρα πολλά προ... υπαρκτά προβλήματα αντιμετωπίζονται ως ε, ταμπού και έτσι δεν βοηθά κανείς, το να τα Αυτό πιστεύω είναι το λάθος του οργανισμού αυτού, που γίνεται λόγος για ρατσιστικές ενέργειες και όλα μπαίνουν στο ίδιο καζάνι. η δημοκρατική νόμιμη πολιτική, ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κόμμα δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στο ίδιο ε, καζάνι με τη ρατσιστική βία. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο οργανισμός ε, αυτός πραγματικά έχει ξεπεράσει το όριο των αρμοδιοτήτων του. Δεν είναι πολιτικά ουδέτερος. Και δεν θα έπρεπε να επιτίθεται σε κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και έχουν και αντιπροσώπους μάλιστα στο Κοινοβούλιο. Κύριε Μπερζέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είχα πρόθεση να παρέμβω, αλλά αφού ορισμένους συναδέλφους αποφάσισα να λάβω το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό για την εργασία του, διότι πιστεύω ότι είναι πολύτιμη για μας σε σχέση με αυτά που μπορούμε να ε, προτείνουμε έμπρακτα και εκπλήσουμε, όταν ε, ζητούν ορισμένοι συνάδελφοι να υποβάλλετε πολιτικής υφής προτάσεις γιατί έχετε τη δυνατότητα προβλέψεων αλλά στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων και της λειτουργίας τους γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα προβλήματα, πού υπάρχει αδιέξοδο και ποιος δεν θέλει να προωθήσει τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε τα πράγματα γνωρίζοντας, γιατί γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη φέρουν την ευθύνη και ιδιαίτερα εκείνα τα οποία δεν θέλουν να προχωρήσουν και αυτό φαίνεται και από τις δικές σας διαπιστώσεις, οι οποίες είναι ε, αρκετά αντικειμενικές. Μας μιλάτε για ορισμένα ε, ζητήματα, μας προειδοποιείτε και θα ήθελα και εγώ να σταθώ στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μίτσελ. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στους κανόνες που υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν ε, ολιστήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης μας το λέει, εσείς μας το λέτε, το είπε και ο Έλληνα συνάδελφος Μας το είπε και ο ειδικό ηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε λοιπόν ε, σε αυτό το σημείο. Ινοβατούν. Μιλάμε για ε, δημοκρατική νομιμότητα. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το ουγγρικό ζήτημα και δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχει δημοκρατική ε, νομιμότητα τότε ε, ξεφεύγουμε και ε, αποτρέπουμε ορισμένα ζητήματα. Θα πρέπει αυτές οι αξίες πραγματικά να εφαρμόζονται στο, στο ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό το δείχνουν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το λέω σε σχέση με τον ε, τελευταίο προλαλήσαντα, η δημοκρατική νομότητα δεν επιτρέπει την προτροπή ε, σε ρατσιστικές δραστηριότητες. Αυτό το είδαμε και με την άρση της ασυλίας της, ασυλίας της κυρίας Λεπέν. Ας αφήσουμε αυτό το έργο στη δικαιοσύνη να κρίνει την κατάσταση. Εάν δεν εφαρμόσουμε τους κανόνες τότε είναι απόλυτα λογικό να μας σύρουν ενώπιον των δικαστηρίων και θα αποαφανθεί η δικαιοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν κόμματα τα οποία έχουν εκλεγεί δημοκρατικά που ξεπερνούν την ε, κόκκινη γραμμή και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όταν μιλάμε εν ονόματι της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω τώρα από τους επισκέπτες μας να απαντήσουν. Να προσθέσω όμως και κάτι που έχει σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ιδιαίτερα με τον τρόπο που υποδέχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όταν φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκεφτήκαμε τη Σουηδία πολύ πρόσφατα, ε, όπου υπάρχει μεγάλη γενεοδορία, κοινωνική γενεοδορία. Αλλά, ωστόσο, μας ανησυχεί το γεγονός ε, ότι υπάρχει μια νέα τάση που παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός παιδιών τα οποία χρησιμοποιούνται από ορισμένου εγκληματίε και καταπατούνται τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους όταν μετακινούνται αυτά τα παιδιά αυτοί οι ανήλικοι από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το συμφέρον τους ε, ως γνώμονα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχουν ε, μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα νομικής ε, προσφυγής. Κάποιον, αν υπάρχουν ένδικα μέσα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρω πως είναι πολλές ερωτήσεις και θα μας τελειώσει ο χρόνος. Ήδη μας έχει τελειώσει ο χρόνος, ωστόσο όμως παρακαλώ απαντήστε. Έχετε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για όλες τις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον Μόρτεν Κέρουμ για να σας απαντήσει. Μόρτεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές ερωτήσεις, πολλές καλές και επικοδομητικές ερωτήσεις και σχόλια για την ετήσια έκθεση. Ξέρω πως ε, ενδιαφέρει τους συναντέλφους που βρίσκονται εδώ, διότι η έκθεση αυτή φυσικά θα επηρεάσει και τους τομείς ε, των δραστηριοτήτων μας και τις επόμενες εκδόσεις της έκθεσης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας σύντομα αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε και διμερώς αν θέλετε. Κύριε Βότσον, καταρχάς, όσον αφορά την ετήσια έκθεση και το πώς μπορεί να συνδεθεί με το άρθρο 2, τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε σε σχέση με το άρθρο 2. Καταρχάς να σας πω ότι το άρθρο 2 βρίσκεται και καλύπτει ήδη πάρα πολλά συστατικά στοιχεία μέσω της ε, εντολής του οργανισμού μας. Και αυτό φαίνεται και από τις συζητήσεις εδώ και από τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο. Συζητήσαμε λοιπόν το πώς εμείς ε, από εδώ και στο εξή θα μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο την ετήσια έκθεση έτσι ώστε να αναφέρεται στους τομείς που είπατε. Πιστεύω πως ο οργανισμός μας μπορεί να συνεισφέρει με γνώση και για τις δικέ μας έρευνες και για το έργο των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα, και, άργο, και άλλων οργανισμών. Να πολλαπλασιάσει τις γνώσεις μας δηλαδή. Υπάρχει τώρα η δυνατότητα του συμβουλίου, στο, Συμβούλιο βασισμένο σε μία δήλωση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός το Συμβούλιο να ζητήσει τη βοήθεια του οργανισμού με βάση το άρθρο 7. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες για διευρυμένες αρμοδιότητες που θα καλύψουν τους ε, τομείς που αναφέρατε και θα πηγαίνουν πέρα από την εντολή μας. Τώρα, όσον αφορά την ε, διάκριση, τις διακρίσεις προς τους ε, Ρώσους της χώρας της Φαλτικής, να πω ότι η έρευνα που κάναμε το 2008 και 2009 μας έδωσε αφορμή να αποφασίσουμε να την επαναλάβουμε και να επαναλαμβάνουμε την ε, έρευνα και τη μελέτη αυτή κάθε πέντε χρόνια. Του χρόνου θα επαναληφθεί λοιπόν αυτή η μελέτη, όχι μόνο για να δώσουμε ένα στιγμιότυπο της εκατάστασης, αλλά και να δούμε τις τάσεις και το πώς αυτές αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου για να δούμε αν οι πρωτοβουλίες, ε, οι νομοθετικές έχουν αντίκτυπο στην μάχη κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, ναι, θα καλυφθεί η ρωσική μειονότητα. Επίσης, όπως αναφέρετε εσείς, εμείς θα συνεργαστούμε στενά και με την Ελίθουανική Προεδρία. Το επόμενο τήσιο συνέδριό μας ε, θα έχει ως θέμα τα εγκλήματα μίσους. Δεν ξέρω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες ε, για τα θέματα του συνεδρίου, πάντως θα καλύπτεται. Τώρα, κύριε Παπα-Νικολάου. όσον αφορά το πώς μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει συζητηθεί στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης, αλλά και στα πλαίσια άλλων δραστηριοτήτων μας. Έχουμε συζητήσει το πώς μπορούμε να οξύνουμε λίγο τις εκθέσεις μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να σας δώσουμε, όπως είπατε, απτές προτάσεις και διαφορετικές ε, επιλογές. Φυσικά υπάρχουν λεπτές ισορροπίες. Δικό σας έργο είναι η χάραξη πολιτικής και εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι βοήθεια γι' αυτό. Όμως ε, γενικά μπορώ να πω ότι τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας μας εμείς ε, δαπανίσαμε πολλά κονδύλια έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για το πώς μπορούμε να καταρτήσουμε τη βέλτιστη δυνατή ετήσια έκθεση. Επίσης, μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα και με τον ε, ειδικό συγγήτη για την μετανάστευση, ασκούμε συντονιστικό έργο. Ήρθε ο ειδικό ε, απεσταλμένος στην Βιέννη και συζήτησε με τους συναδέλφους μας, είδε τη δουλειά που κάνουμε, ιδιαίτερα στο θέμα των ελληνοτουρκικών ε, συνόρων. Υπάρχει, μπορώ να πω, μία ολαιόνα και, και... και αυξανόμενη ενισχυμένη συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων. Και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος υπήρχε εξαιρετική συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τα εγκλήματα μίσου, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουμε μαζί με την Eurojust, Justin Seapol και την Ευρωπόλ για να δούμε τι μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας από εμάς έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα μίσους και να έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών έτσι ώστε να συνεργαστούμε καλύτερα. Τώρα, κυρία Στανόκα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, συλλογή δεδομένων. Αυτό που ελπίζουμε να καταφέρουμε, για παράδειγμα ε, με τη δουλειά που κάνουμε τώρα πάνω στους ε, Ρωμά, συνεργαζόμαστε με 12 κράτη-μέλη, να σας πω, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε ορισμένους βασικούς δείκτες, τους οποίους μπορούν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, αφορώντας εθνικούς μηχανισμούς παρακολούθησης. Ελπίζουμε αυτό να είναι μια όθηση για να προχωρήσουν για να προχωρήσει η μάχη όχι μόνο για την διάκριση κατά των Ρωμά αλλά και άλλων ομάδων. Όπως σας είπα, είμαστε πέντε χρόνια ως οργανισμός και ακόμα αναπτυσσόμαστε. Αλλά ελπίζω η δουλειά που έχουμε κάνει με τους Ρωμά να διοχετευθεί μέσω καλών πρακτικών και σε άλλους τομείς. Όπως είπα, απαντώντας επίσης την προηγούμενη ερώτηση για τα εγκλήματα μίσους, και εδώ συνεργαζόμαστε μαζί με την Ευρωπόλ, την Eurojust και άλλες υπηρεσίες για να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία πάνω σε δύο ή τρία βασικά σημεία για να ελέγξουμε τα εγκλήματα μίσους και να τα αντιμετωπίσουμε και να τα χωρίσουμε είτε σε περιπτώσεις ε, απλής βίας είτε σε περιπτώσεις ε, δολοφονιών. Αυτό πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πάρα πολύ διότι δεν έχουμε μόνο τα στοιχεία αυτά από τις τέσσερις χώρες τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε αυτές ε, τις χώρες όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Διότι μας λείπουν πολλά ακόμα. Αλλά φέτος θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα εγκλήματα μίσους και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα κύριε Μπρόντς, όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, Φυσικά όλοι είμαστε υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του λόγου. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει κεφάλαιο σε αυτό που αναφέρατε είναι ότι δεν είναι κομμάτι των αρμοδιοτήτων μας. Όπως θα δείτε, εμείς ακολουθούμε ένα γενικότερο πλαίσιο. Επίσης θα δείτε ότι όλα αυτά που κάνουμε πάνω στα εγκλήματα μίσους ε, δεν εστιάζονται στην ρητορική μίσους. Εστιαζόμαστε μόνο στα εγκλήματα μίσους. Να σας ε, διαβεβαιώσω όμως ότι πραγματικά μας ε, απασχολεί πάρα πολύ η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της. Και φυσικά ασχολούμαστε και με την διάσταση της ρητορικής μίσους. Διότι πολλές φορές είναι ένας πρόδρομος των εγκλημάτων μίσους. Τώρα, κυρία Μέτσολα, Μάλτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και που έχουμε κάνει μέσω διαφόρων εκδόσεων είναι να αυξήσουμε την αλληλεγγύη. Και την αλληλεγγύη μάλιστα ως ένα από τα συστατικά στοιχεία της ε, προστασίας. Και αν δούμε την ιστορία, τη μεταναστευτική ιστορία και την προστασία των μεταναστών, θα δούμε ότι η αλληλεγγύη είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό στοιχείο όσον αφορά τους πρόσφυγες. Είναι αναγκαία η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και είναι δυνατόν. Το, 1979, να σας θυμίσω, είχε διεξαχθεί το συνέδριο στην Γενέβη όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν μέτρα για τους 250.000 πρόσφυγες από το Βιετνάμ. Πιστεύω πως ε, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, κύριε Κλέης, πάλι για την ελευθερία της έκφρασης και την ε, δημοκρατική νομιμότητα, να σας πω ότι Φυσικά και δεν αμφισβητούμε την δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό όμως που αμφισβητούμε και που συζητούμε είναι ανεξάρτητα από κομματικές αποχρώσεις, κύριο μέλημά μας είναι να δούμε το πώς θα προστατεύσουμε τις μειονότητες. Και πώς αυτό θα γίνει πράξη και πώς αυτό θα μεταφερθεί σε πολιτικές ενέργειες. Αυτό κάνουμε. Ολοκληρώνω σε λίγο. Κυρία Βερζιά. πιο πολύ σχόλιο ήταν αυτό που κάνατε, αλλά αναφερθήκατε στο άρθρο 2 και τις αξίες του άρθρου 2. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους και το πώς χρησιμοποιούνται από εγκληματίες. Ε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι φυσικά με τα στοιχεία που έχουμε στην έκθεσή μας από το 2009, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους και την διακίνηση παιδιών, πρόκειψε ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών, τα οποία βρίσκονταν σε κέντρα υποδοχής ετούντων άσυλο, τα οποία ε, στην αρχή καταγράφηκαν και μετά εξαφανίστηκαν είτε μέσω παράνομων υιοθεσιών, είτε μέσω ε, της ε, βιομηχανίας ε, πορνείας, είτε μέσω δωρεών οργάνων εντό εισαγωγικών. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε, αυτήν την, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όντως δεν υπάρχουν ακόμα τα κατάλληλα συστήματα, οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να προστατευτούν τα παιδιά. Για τον οργανισμό μας φέτος, μεγάλο βάρος έχει η σκλαβιά, η δουλεία και οι ακραίες μορφές εκμετάλλευσης στην αγορά εργασίας. Και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαίτερη μνήμα στα παιδιά στην ε, μελέτη αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι είμαστε ευγνώμονε που ήρθατε σήμερα και μας μιλήσατε και παρουσιάσατε την έκθεσή σας και παρουσιάσατε αναλυτικά τα θέματα και δώσατε εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την επίσκεψη στη Βιέννη σε άλλο σημείο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σα ευχαριστώ και του δύο. Uh, um, για το σημείο 4 ζήτησε ο Πρόεδρος μια και είναι σχετικό θέμα, είναι παρουσίαση της εκθέσεως για την αντιπροσωπεία που επισκέφθη με τον οργανισμό, επισκέφθηκε τον οργανισμό το Φεβρουάριο. Επικεφαλής ήταν ο πρόεδρός μας. Αποτελείται από τις αδερφούς τον κύριο Παπα-Νικολάου και την κυρία Τζανόκα και η κυρία Λούνατσεκ ήταν συνόδευση επιτόπου τη εργασία ντόπιο μέλος. Στόχος αντιπροσωπεία είναι να γίνει δελεχή ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τι αδικέ προτεραιότητε του οργανισμού για το 2013 και περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις νομοθετικές και νομοθετικές διαδικασίες και βοήθεια που θα δώσει ο οργανισμός στο Κοινοβούλιο εν ώψη του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2013-2017. Συναντήθηκε η προσωπία με το διευθυντή της οργανισμού, τις επικεφαλής, τους ματάρχες, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους με κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που εργάζονται εντό του φορέα. Διάφοροι εμπειρογνώμονε παρουσίασαν λεπτομερώ ε, τα πιο πρόσφατα προγράμματα, σχετικά προγράμματα του οργανισμού και τρει έρευνε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βία κατά των γυναικών, εμπειρία που έχουν οι ΛΟΑΤ και ποια είναι η κατάσταση των ε, κοινοτήτων των Εβραίων. Και καλύφθησαν εννέα χώρε, οργανισμού και μέσα στην αντιπροσωπεία για απορίσματα την έρευνά τη για την αντιμετώπιση των μεταναστών που καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εξωτερικά σύνορα αυτή. Η αντιπροσωπεία τόνισε την ανάγκη ο οργανισμό να επαναλάβει τακτικά τι εκθέσει αυτέ και τι έρευνε για να εντοπίσει τη στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να κρούει τον κόσμο του κινδύνου όταν αντιμετωπίζονται κρίσει, να βλέπει κατά πόσο υπάρχουν κίνδυνοι εξτρεμισμού στην Ευρώπη και θα πρέπει να αναφέρει τι καλέ πρακτικέ στα διάφορα κράτη-μέλη και να δίνει πιο συστηματική νομοθετική λύση όσον αφορά την πολιτική και προτάσει για πολιτική βάση στοιχείων. Κάποιε δράσει συνεχείας συζητηθήκαν, κυρίω να υπάρχει συμβουλή εμπειρογνωμόνων, συγκεκριμένο στόχο από τον οργανισμό, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και διαδικασίες ε, ασύλου, προστασία των δεδομένων, διακριτική μεταχείριση και όπως ανέφερε και ο μιλητής την ένταξη των Ρωμά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει ενδεχόμενο ρόλο του οργανισμού για να παρακολουθεί τα θέματα εξτραμιστικών ομιλιών και ε, ομιλιών μίσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελευταία συζήτηση αφορούσε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους αυστριακών μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων φορέων σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο σημείο. Αυτά μου ζήτησα να σας πω, Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλετε, όσοι ήσασταν παριστάμενοι σε αυτήν την αντιπροσωπεία, να θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Εν συντομία, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ζητήστε το λόγο. Αλλιώς θα προχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 5 κυρίες και κύριοι. Αν έχετε την καλοσύνη πάμε εκεί. Η απελευθέρωση του δυναμικού α, ε, α, της, ε, της χρήσης του cloud computing στην Ευρώπη η συγγητρία είναι η κυρία Τζούθης Αργεντίνη των Πρασίνων στις 29 Μαΐου στην Επιτροπή Ελευθεριών παρουσιάστηκε σχέδιο γνωμοδότησης από πλευράς Τζουντίθ Έκτοτε 54 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και μετά ε, θα ξεκινήσουμε συζήτηση με τα μέλη και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω ότι θα προβεί σε κάποια σχόλια σχετικά με τις υποβληθείς τροπολογίες. Λοιπόν, Τζούντιθ, παρακαλώ. Τόση μεγάλη χαρά να σας βλέπω στη θέση του Προέδρου. Ευχαριστώ. Όλοι κινούμεθα προς το θέρος. Δεν ξέρω αν οι παρίστανται για να σχολιάσουν. Πέρα από τις 54 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, είχαμε και το πρόβλημα του πρίσμ και το τεμπόρα, δύο σκάνδαλα που άλλαξαν εν μία νυχτή τη συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων και συλλογής δεδομένων. Νομίζω ότι θα αλλάξει και κάπως η άποψη της εκθέσεως για τους υπολογιστές, το υπολογιστικό νέφος. Εγώ όπως και κάποιοι σκιώδεις ε, έχουμε υποβάλει τροπολογίες που διευκρινίζουν την κατάσταση. Λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας όχι μόνο κατά των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο αλλά και έναντι ενδεχομένων τρίτων χωρών, καθώς και έναντι των κυβερνήσεών μας. Και παροτρύνουμε το θέμα αυτό να εξεταστεί για τη συλλογή των στοιχείων. Έχω διανύμει ήδη σχέδια κειμένου, συμβιβαστικές τροπολογίες μάλλον προς τους συναδέλφους, από τις 54 τροπολογίες που υπευλήθησαν οι περισσότερες είναι πολύ επικοδομητικές και θα προσπαθήσω να τις συμπεριλάβω σε συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που μοιάζουν και έχουν παρόμοιο υπόβαθρο. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας, κατά πόσο έχω ήδη καταφέρει να συμπεριλάβω τις σκέψεις σας στις συμβαστικές τροπολογίες ή αν αισθάνεστε ότι έχετε μείνει εκτός θα δώσω τις τελικές συμβαστικές τροπολογίες μετά τις θερινές διακοπές. Όμως υπάρχει μια τροπολογία, η τροπολογία 45 ε, του κυρίου και της κυρίας Γκάμπριελ που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ θα έλεγα να μην να μην συμπεριληφθεί αυτό το τμήμα διότι αντιβαίνει των επιχειρημάτων μου. Εγώ ζητώ διαφάνεια, ανοιχτή προσέγγιση και προστασία πολιτών. Οπότε ερχόμαστε πίσω στο θέμα της άκτα που καταψήφισε το Κοινοβούλιο. Έχουμε δύο τροπολογίες που θα ήθελα να διευκρινιστούν. Την 46 του Μάρκο Σκούρια και 47 του Λορέντσο Φοντάνα που θέλουν να δοθεί προσοχή στους ευάλωτους χρήστες και στην προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Πώς να το ερμηνεύσω αυτό, αν είναι παρόντες οι συνάδελφοι να μου εξηγήσουν. Αλλιώς ίσως μπορείτε να συνειδητοποιήσετε να μου στείλουν απαντήσεις. Πώς να ερμηνεύσω αυτές τις τροπολογίες να ξανασκεφτώ την συζήτηση που είχαμε για την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στο διαδίκτυο, εκμετάλλευση των παιδιών και αν ναι, πώς μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε την γνωμοδότηση. Αυτά είναι τα σχόλια που έχω για την ώρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους Κιώδης τους παρόντες να συμβάλλουν στη συζήτηση. Ο Άξελ Βος είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία, καταρχάς όσον αφορά τις τροπολογίες. Να η τροπολογία 28 της κυρίας Σιντφέλντ με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνα, τη θεωρώ πολύ καλή και πιστεύω πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπεριληφθεί, ακριβώς όπως και η τροπολογία 23 της κυρίας Χάνκες. Ωστόσο, αυτό που θεωρώ περιττό είναι η τροπολογία 13 της εισηγήτριας και η τροπολογία 36 της κυρίας Ζίπελ. Διότι οι ρυθμίσεις αυτές τις οποίες αναφέρονται πιστεύω πως ε, είναι αυτονόητες. Και θα έπρεπε να βρίσκονται στον κανονισμό. Και όχι εμείς να κάνουμε κάτι πάλι καινούριο και να το αναφέρουμε από την αρχή. Κάτι που ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση της εισηγήτριας για την τροπολογία 46 να σας πω ότι και εδώ ε, είναι μια τροπολογία που πιστεύω πως ταιριάζει στον κανονισμό και όχι στην έκθεση. Πιστεύω ότι εδώ αυτή η έκθεση είναι σημείο ε, στο οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε την προστασία δεδομένων και τίποτα άλλο. Τώρα, τροπολογία 2. Τι θεωρώ εντάξει. Όσον αφορά την τροπολογία 21 και την τροπολογία 26, εδώ θα ήθελα μια καλύτερη διάκριση για λόγους ταξινόμησης και τώρα στην τροπολογία 43 πιστεύω ότι επίσης είναι αυτονόητο αυτό που αναφέρεται για αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω πως είναι τόσο αυτονόητο, ώστε δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται και εδώ. Είναι κάτι που αναφέρεται ως σε δικαίωμα. Αυτά προς το παρόν από μένα. Ε, η τροπολογία 53 πιστεύω πως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί. Τώρα όσο για την τροπολογία 48 να πω ότι δεν νομίζω πως έχει διατυπωθεί σωστά. Εγώ προσωπικά βρίσκω τη δική μου πρόταση καλύτερη. Όσον τώρα αφορά τις εμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκε η συγγήτρια ιδιαίτερα την 4α και την 2α, να πω ότι αυτές είναι καινούριε. Η 4α αναφέρεται στο, στο θέμα της κατασκοπίας και στο πρόγραμμα PRISM. Στην Ολομέλεια ψηφίσαμε και εγκρίναμε ένα ψήφισμα και πιστεύω πως δεν χρειάζεται άλλη μία φορά να αναφερόμαστε σε αυτό στο κείμενο. να αναφερθούμε στους ε, λόγους, αλλά πιστεύω πως θα ήταν υπερβολικό να αναφερθούμε πάλι από την αρχή. Το μπορούμε να αναφέρουμε το ψήφισμα της Ολομέλειας και να το σεβαστούμε. Τώρα, το 2α, η νέα. Και εδώ βρίσκω ότι ο κανονισμός είναι το καλύτερο μέρος για να βρίσκεται κάτι τέτοιο και όχι έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζήπελη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ στις ε, επιμέρους τροπολογίες, αλλά να πω κάτι βασισμένο σε αυτά που είπε ο κύριος Φως. Ναι, ορισμένα πράγματα ενδεχομένω είναι αυτονόητα. Αλλά, εάν διαγράφαμε από, το, από την νομοθεσία μας όλα αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε αυτονόητα, τότε σίγουρα τα κείμενα που θα είχαμε θα ήταν πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο μικρά. Πιστεύω πως δεν πειράζει, δεν κάνει κακό να αναφέρονται ξανά κάποια πράγματα, τον συνδέονται μεταξύ τους, γιατί αν κάποιος θεωρεί κάτι αυτονόητο δεν σημαίνει ότι το θεωρούν όλοι αυτονόητο. Επίσης, όσον αφορά τις κυρώσεις, Παρομοίω, δεν θεωρώ υπερβολικό να αναφερθούμε ξανά στι κυρώσει, γιατί το σύστημα υπολογιστικού νέφου είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει μέχρι τώρα. Τώρα, όσον αφορά το πού θα βρίσκεται αυτό το υπολογιστικό νέφο, υπάρχουν ορισμένοι πάροχοι οι οποίοι δεν έχουν ένα μόνο χώρο, αλλά πολλούς και εκεί και αποθηκεύουν λοιπόν τα δεδομένα του νεφού σε, πολλούς, ε, σε πολλές ε, τοποθεσίες, έτσι ώστε αν ε, πάθει κάτι ο ένα σερβερ να μεταφέρονται στον άλλο και γι' αυτό πιστεύω ότι οι κυρώσεις πρέπει να αναφέρονται ρητά. Τώρα όσον αφορά το πρίσμ και αν είναι επίκαιρο μια που το ψηφίσαμε στην Ολομέλεια, ναι, έχουμε ένα ψήφισμα μένα από την Ολομέλεια. Αυτό δεν αποτελεί όμως ε, διαπραγματευτική βάση. Υπάρχει εδώ μια άλλη διάσταση, την οποία πρέπει να τονίσουμε, διότι δεν αφορά μόνο την προστασία δεδομένων. Διότι οι μυστικές υπηρεσίες υπόκειται σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να σκεφτούμε καινούριου νόμους για τα νέα προϊόντα τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να μην έχουν οι μυστικές υπηρεσίες πρόσβαση χωρίς καμία νομοθετική ρύθμιση σε αυτά τα νέα προϊόντα. Το υπολογιστικό νέφος είναι ένα από αυτά τα νέα προϊόντα το πρόβλημα εδώ δεν είναι η προστασία των δεδομένων, αλλά και σε αυτό και στα άλλα προγράμματα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ε, πολλά κράτη-μέλη τα οποία θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να έχουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να τονίσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και την προσπάθεια να συμπεριλάβει τις προτάσεις όλων μας. Πιστεύω ότι το θέμα του υπολογιστικού νέφους είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να τονίσουμε πώς έχει η κατάσταση, τι είναι αυτό που θέλουμε και να μας δώσει μια καλή αφορμή και αφετηρία να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες του υπολογιστικού νέφους για να ασχοληθούμε με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Όπως ανέφερε γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα υπό το φως του σκανδάλου Πρίσμ και των όσων συμβαίνουν. Συμφωνώ με την κυρία Σίπελ όσον αφορά την προσέγγιση, όπως την εξήγησε. Όσον αφορά στις αστικές τροπολογίες, εν γέννη συμφωνώ με αυτές, διότι θεωρώ ότι καλύπτουν τις ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κινδύνους από το υπολογιστικό νέφος για τους χρήστες. Χαίρομαι διότι βλέπω μια πληρέστατη παράγραφο όσον αφορά τα προβλήματα της παρακολούθησης μεγάλης κλίμακας από ξένες αρχές. Και αν ακόμα δεν υπάρχει προφανής λύση, θα πρέπει να αναφέρεται σαφέστατα κάτι που προτάθηκε στις τροπολογίες που υπέβαλαν κάποιοι συνάδελφοι και εγώ. Είχα συμπεριλάβει έτσι και μία πρόταση να ζητάμε από εταιρείε υπό τη δικαιοσία τρίτων χωρών να παρέχουν στους χρήστες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφή προειδοποίηση όσον αφορά την πιθανότητα τα στοιχεία τους ίσως να υπόκεινται σε παρακολούθηση από τις αρχές τρίτων χωρών και χαίρομαι που βλέπω ότι η Σοφή Ιντβελτ ζήτησε κάτι παρόμοιο. Εν ώψη των νέων εξελίξεων ίσως υποβάλλουμε και άλλες τροπολογίες. Εν γέννη όμως πιστεύουμε ότι η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι σύντομη και να περιέχει τις προτεραιότητες μας. Τερίες προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ζητήσω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Η κυρία Βαντέκα. Sorry, one of you... Κάποιος από εσάς. Ζητώ συγγνώμη, η κυρία Βαντέκα, η συνάδελφός μου δεν είναι εδώ. Τσάλβος είμαι. Μιλάω από DG Connect. Έγινε συνεδρίαση. Συνομιλία με την ε, Επιτροφή σας, ο κ. Καμπαλάρο, ο κ. Μαντέους μίλησαν, συνάδελφοί μου μίλησαν τότε. Ισχύουν αυτά που υπόθηκαν και τότε και τώρα. Μπορώ να επαναλάβω αυτές τις απόψεις. Κατά λοιπά, να δώσω στους συναδέλφους Didi Just το λόγο, διότι πολλά από αυτά που αναφέρονται, οι παράγραφοι της γνωμοδοτήσεως, αφορούν προστασία δεδομένων. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε συγκεκριμένα σχόλια όσον αφορά τις τροπολογίες. Χαιρόμαστε με τα αποτελέσματα που πετέχθησαν στις συζητήσεις. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, η συγγήτρια. Η κυρία Σίπελ ε, το είπε πολύ εύκολα ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει τίποτα που να θεωρείται αυτονόητο. Πολλοί θεωρούν αυτονόητο ότι τα στοιχεία στο ε, νέφος χρήζουν προστασίας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό αυτή τη νέα τεχνολογία και τον νέο τρόπο εργασίας που θα αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη ως προς τη μεταχείριση των δεδομένων για να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα. Βεβαίως, αν πρέπει αυτό να γίνει, έχει καλώς Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναθεωρούμε τις θέσεις μας από καιρού εις καιρόν, διότι έξι μήνες πριν ποτέ δεν θα θεωρούσαμε ότι το υπολογιστικό νέφος είναι τόσο σημαντικό όσο το θεωρούμε τώρα. Ε, προωθούμε νέες προσεγγίσεις και προσαρμοζόμαστε με την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο θα δω το ψήφισμα της προηγούμενης εβδομάδας για να δω κατά πόσο συμβαδίζουμε. Όχι για να βγάλουμε αυτά που ενυπάρχουν, αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι ε, δεν υπάρχει διχασμός μεταξύ των δύο. Ως πως περισσότερες τροπολογίες κύριε Τρενταφυλλίδη ε, έχει ε, έχουμε περάσει αυτό το σημείο, αλλά πιο ξέρει κάτι μπορούμε να κάνουμε με προτάσεις συμβιβασμού. Πρόεδρος, ως προς τις ημερομηνίες θα ψηφίσουμε στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στη συνάντηση αυτής της Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε την εκθέση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 5 αρχίζουν οι ψηφοφορίες, γι' αυτό θα ήθελα όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν με τις κάρτες τους. Στις 5 λοιπόν. Σημείο 6 της ημερήσιας ε, διάταξης που είναι ο προπολογισμός του 2014. Ο Γιάννη Μιλντερ είναι ο εισηγητής, αλλά η Σόφη θα παρουσιάσει το θέμα εξ ονόματός του. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τα γενικά στοιχεία του προϋπολογισμού που σχετίζονται με την Επιτροπή μας και μετά θα ε, εισηγηθεί η Σόφη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το σχέδιο προϋπολογισμού 2014. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τα συμφραζόμενα εργασίας και τους περιορισμούς μας στη μέθοδο εργασίας. Νομίζω ότι σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όπως και πέρυσι αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού συντάχθηκε στα πλαίσια δημοσιονομικής λιτότητας με οροφές και μειώσεις στο προσωπικό που γνωρίζουμε ότι απορρέουν από την οικονομική κατάσταση. Πέρα όμως από αυτά τα συμφραζόμενα υπάρχει και κάτι διάζων που θα πρέπει να αναφερθεί. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι το οποίο ε, έχει δυσκεράνει την κατάσταση. Επειδή πρόκειται λοιπόν για το πολιετές πρωτίστως, οι προτάσεις επιτάπητος λαμβάνουν υπόψη την ε, προχωρημένη συζήτηση ως προς το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του Ιουνίου του 2013. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή ανακύψει με βάση τις προσαρμογές θα ενταχθεί στον προπολογισμό με διορθωτικές επιστολές στο σχέδιο προπολογισμού τέσσερα ε, στάδια. Αυτό, αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να σας δώσω. Ως προς την νομική βάση, επειδή μιλάμε για άσυλο και μετανάστευση και το Ταμείο ως προς την εσωτερική ασφάλεια, ε, στα πλαίσια της Γενικής ε, Διεύθυνσης Home Affairs και μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης και δικαιωμάτων και εσωτερικών υποθέσεων και σχετικής Γενικής Διεύθυνσης Γνωρίζετε ότι η νέα νομική βάση έχει τεθεί υπό συζήτηση και θα μπορούσαμε να, μάλλον θα πρέπει να διευθετήσουμε και άλλα θέματα ως προς την προχρηματοδότηση, την πολιετή προχρηματοδότηση. Όσον αφορά την ε, τυπολογία που, μας, ε, που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα, με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής για την ονοματολογία θα προτείνουμε κάτι με μεγαλύτερη διαφάνεια και στοχοθετημένο. Αυτό έγινε και αντικατοπτρίζει τους ειδικού στόχους της νέας νομικής βάσης και θεωρούμε ότι είναι θετική η εξέλιξη. Εξάλλου, ως προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, λαμβάνουμε υπόψη τα items του προϋπολογισμού που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα. Με βάση αυτό το γενικό πλαίσιο τώρα μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες ιδιαίτερα ως προς την ασφάλεια και την ηθαγένεια, δηλαδή κεφάλαιο 3 σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων για το νέο ταμείο, το ποσό που προτείνει η Επιτροπή αντικατοπτρίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως έχει προσαρμοστεί μετά από τις υποδείξεις του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου και που δέχτηκε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 26 ε, Ιουνίου του 2013. Για το 14-20 η Συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου προβλέπει μία μείωση του 16,6% και αυτό θα ισχύσει για το 13 και το 14. Τώρα, ως προς τις πιστώσεις πληρωμών, ήμασταν ιδιαίτερα σύνετοι γιατί θέλουμε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νέα προγράμματα με βάση τον ελάχιστο αυτό παρονομαστή, ιδιαίτερα για το 14. Ίσως εγκρίνουμε αργά τα κονδύλια και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και έτσι έχουμε μερική χρηματοδότηση του πλαισίου προχρηματοδότησης του 14 ως προς την αρχική προγενέστερη χρηματοδότηση, προχρηματοδότηση που είναι υποδιαπραγμάτευση θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις πιστώσεις υποχρεώσεων του 2014. Τώρα ως προς τους οργανισμούς. Η πρόταση της Επιτροπής διέπεται από δύο βασικές δεσμεύσεις, το, τις ενδεικτικές δαπάνες, αναθέσει μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τον στόχο μείωσης του προσωπικού στον οργανισμό της τάξης του 5% μέσα σε μία πενταετία. Επιπλέον η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πλήρωση θέσεων προσωπικού με φάση ε, τα, τις νέες δραστηριότητες για τους οργανισμούς που, έχουν, ε, που ήδη λειτουργούν εδώ και χρόνια θα γίνει ένα πάγωμα το 14, στάξη του 7,14 εκτός από τους οργανισμούς που, θε, που εντάσσονται μέσα, μέσα στα νέα καθήκοντα, δηλαδή τη Frontex. Η Επιτροπή έχει διαφορετική προσέγγιση για τους οργανισμούς που θεωρούνται startups, δηλαδή η Ιουλίζα και Άζο, γιατί έτσι θα μπορέσουν να έχουν επιπρόσθετους πόρους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Τέλος, Πρόεδρε, η συνολική συνεισφορά για τις αποκεντρωμένους οργανισμούς στη θέση 3 το 14 αποτελεί αύξηση, παρουσιάζει αύξηση του, της τάξης 4,9% αν συγκρίνουμε το 13. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η αύξηση απορρέει από τη την ε, ε, θέση λειτουργία του οργανισμού EU LISA ε, ελπίζω αυτές οι διευκρινήσεις να ήταν ε, σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα η Σοφή Ιντβέλτ να παρουσιάσει την, τις δικές της Θα σας διαβάσω μια δήλωση. Ο συνάδελφος ε, ζητά συγγνώμη γιατί δεν είναι παρόν και βρίσκεται αλλού, έχει μια αποστολή και ακόμα και ο Γιάννου Μούλτερ δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Στις 26 Ιουνίου η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού 14. Ο, ως εισηγητής της ΛΥΜΠ, ο Γιάννου Μούλτερ προτείνει τα εξή και λέει τα εξή λυπάται για τη μείωση του 9,4 και 8,3 αντιστοίχως σε υποχρεώσεις ε, σε δαπάνες, ε, σε υποχρεώσεις και πληρωμές. Και λυπάται διότι η νομική βάση ε, την χάνει διαπραγμάτευσης. Ο Γιάνν Μίλτερ τάσεται υπέρ της ιδέας ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να απορροφηθεί. Τα τέσσερα κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τη συνεργασία εκεί όπου υπάρχει Υπάρχουν κοινά καθήκοντα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία για το άσυλο και τη μετανάστευση και θα πρέπει να υπάρξει επαρκή συνεισφορά από τα κράτη-μέλη. Ο Μίλτερ πιστεύει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προγράμματα τα οποία πρόσφατα έχουν εγκριθεί. Ευχαριστώ. πολύ. Κύριε Κέλλερ, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και την Σοφή Ινφέλντ. Το σχέδιο γνωμοδότησης που έχουμε είναι κάτι το οποίο βρίσκω εξαιρετικό, ιδιαίτερα το σημείο 2, το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όντως είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού όταν δεν έχουμε δηλώσει από το Συμβούλιο πώς να κάνουμε τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν. Έχω δύο σχόλια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταρχά, πιστεύω ότι στο σημείο 3 πρέπει επίσης να αναφερθεί η αναγκαιότητα του να υπάρχει προστιθέμενη αξία για τα κονδύλια που να δαπανώνται εδώ. Γιατί πολλές φορές φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια για πράγματα τα οποία θα έκαναν έτσι και αλλιώς, για πράγματα για τα οποία θα δαπανούσαν κονδύλια έτσι και αλλιώς. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε να προστίθεται ευρωπαϊκή αξία στα κονδύλια που διαθέτουμε. Έπειτα, στην παράγραφο 5, δεν είμαι σίγουρη ε, γιατί αναφέρεται ξεχωριστά η Frontex εδώ. Ε, δεν ξέρω επίση αν πρέπει να αναφερθεί η γύρωση, διότι ήταν ένα παράδειγμα κατά το οποίο είχαν ήδη δαπανηθεί κονδύλια, προτού δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα κονδύλια αυτά πριν από ένα μήνα. Γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω πως εδώ είναι καλό να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως προηγούμενο. Και γιατί να πάρει η Frontex περισσότερα χρήματα. Τι γίνεται με την ΕΑΣΟ για παράδειγμα. Έχουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 4. Και εάν θεωρείτε πως είναι μια προτεραιότητά σας, τότε αξίζει να δώσετε και περισσότερα κονδύλια σε αυτήν την υπηρεσία. Και ήδη Frontex λαμβάνει αρκετά από αυτά τα κονδύλια. Αυτά ήταν τα δύο σχολεία μου. Ελπίζω ο εισηγητής να συμφωνήσει. Ευχαριστώ. Κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην ουσία θα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Κολμάιερ. Μιλώ εξ ονόματος λοιπόν της κυρίας Χολμάιερ. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Μούλντερ για μια πρόταση που είναι πολύ καλή. Σημερίζεται τις απόψεις του εισηγητή για το θέμα ως προς την αύξηση του 3 κατά 3% το θεωρεί απαράδεκτο. Ε, ε, θα ήθελε να τονιστεί η σημασία των οργανισμών, ιδιαίτερα των οργανισμών που ε, είναι ιδιαίτερα λειτουργικοί. Η Μόνικα θεωρεί ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στη Europol, όχι μόνο στη Frontex. Και επειδή υπάρχουν, ε, του έχουν ανατεθεί ε, νέα καθήκοντα, δηλαδή την καταπολέμηση του εγκλήματος στον ε, κυβέρνοχώρο. Σε σχέση με τις προτάσεις της κυρίας Χολμάιερ θα ήθελα να πω ότι τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει η αύξηση του προπολογισμού και αυτό όταν εγκριθεί η νομική βάση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πακέτο για τα ευφύ σύνορα και θεωρεί ότι αυτό το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί τάχιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια για το σημείο αυτό από τις άλλες ομάδες ίσως. Θα θέλετε να συνεχίσετε, να πείτε κάτι παραπάνω και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα θέλετε το λόγο, έτσι. Προθεσμία για τις τροπολογίες, 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Εάν η Επιτροπή δεχθεί να γίνουν ε, αποδεκτές τροπολογίες μόνο στην αγγλική γλώσσα, διαφορετικά Προθεσμία για τροπολογιε είναι η 14η Αυγούστου έτσι ώστε να γίνει μετάφραση. Συνήθως αυτό που κάνουμε τέτοιε εποχές είναι να σφίξουμε τα δόντια και να ελπίζουμε να υπάρχουν μόνο τροπολογίες στα αγγλικά, διότι διαφορετικά οι διακοπές μας συρρυκνώνονται. Θα ήθελα λοιπόν να στήσω από την Επιτροπή να δεχτεί τις τροπολογίες μόνο στα αγγλικά έτσι ώστε να τις ε, συζητήσουμε και να τις ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα. Η ψηφοφορία θα αρχίσει ακριβώς στις 5. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε την ψηφοφορία σε ένα λεπτό. Okay, ladies συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ελπίζω να έχετε τι κάρτε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίζω να τι έχετε, υποθέτω πω τι έχετε. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Γέννης Ρόντε ο προτείνω να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Λόγος για την ψηφοφορία είναι ότι η Επιτροπή Ήτρε και ΙΜΚΟ είναι συνυπεύθυνες. Έχετε όλοι τα χαρτιά σας. Αρχίζουμε λοιπόν και παρακαλώ να έχετε υπομονή μαζί μου. Δεν έχω την ταχύτητα που έχει ο πρόεδρός σας, αλλά ελπίζω να είμαστε εντάξει. Καταρχάς, αρχίζουμε. Τροπολογία 60. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. 18 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Τροπολογία 6 υπέρ. Καταπίπτει, συγγνώμη. Η 6 καταπίπτει. Όχι, η τροπολογία 63 είναι αυτή που καταπίπτει. Η γραμματεία μου λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 6. Συμφωνείτε? Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 72. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 21 ψήφι κατά. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Είναι χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 73. Ζήτω συγγνώμη. Τροπολογία 73 είναι χωριστή ψηφορία κατά τμήματα, όπως ζητήθηκε από τους πράσινους. Πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 κατά τμήματα, όπως ζήτησαν οι πράσινοι, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 12. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ, τροπολογία 82. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνατε λοιπόν. Η 83 είναι ταυτόσιμη. Και η 14 περνάμε στην συμβιβαστική 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, υπέρ. Oh, okay. 86. 86, υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 16. Πέρας. Μπορείτε παρακαλώ να σηκώνετε όλοι το χέρι σας. 9 ψήφοι υπέρ 28 κατά Απορρίπτεται σαφώ. Περνάμε στην 89. Ποιο είναι υπέρ. ποιο είναι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 91 παρακαλώ. Πέρας. 15 ψήφοι υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 92, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 93, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίνεται. 19 και 99 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 20. Ψηφίσατε. Πέρας. Πάλι καλά που υπαλληθεύσαμε ηλεκτρονικά. 19 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 και 110 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 και 112 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 28 και 112. Ψηφίσατε. Πέρας. 18 υπέρ 19 κατά. Εκτός μικροφώνου. Ναι, όταν ολοκληρώνεται η ψηφοφορία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σωστά. Τι λέτε. Όχι, δεν δωροδοκούμε. Εκτός μικροφώνου. What does she mean? If colleagues agree, I'm happy to repeat that vote. Θα επαναλάβω την ψηφοφορία αν συμφωνείτε. Ας επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορια τροπολογης τροπολογίας 28-112. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ τώρα και 16 κατά. Κάποιος άλλαξε άποψη λοιπόν. Εγκρίνονται. 113. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται 114. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 115. Πέρας. 16 υπέρ 21 κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 31. Πέρας. 22 υπέρ, 15 κατά. Έγκρινατε λοιπόν. Τροπολογία 32. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 και 118 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. 21 υπέρ, 17 κατά. 34. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος... Αποχές. Δεν βλέπω αρκετά χέρια κυρίες και κύριοι. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 34. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Μάλιστα. Παρακαλώ όλοι ας σηκώσετε τα χέρια σας γιατί κουράζει αυτό. Απορρίπτεται 29 κατά 9 υπέρ. 119. Τις κάνουμε σε μπλοκ 119 μέχρι 122. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 35 παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται 9 υπέρ 28 κατά 123. Ποιος είναι υπέρ. Να τις κάνουμε και αυτές σύνολο λέει ο πρόεδρος. Συμφωνείτε 123 έως 131. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε για την 39 ψηφίσατε όλοι πέρας 22 υπέρ 16 ψήφι κατά εγκρίνεται και άλλη ομαδική ψηφοφορία 133 μέχρι 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά έλεγχος της συμβαστικής 8. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 με 15. Εγκρίνεται. Πάμε στην 142 τώρα. 142 με 144 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 145. Και άλλη ομάδα. 145 μέχρι 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ για τη 43. το ολοι όλοι. Τέλος. 17-21 απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά έλεγχος η τροπολογία 1 ψηφίσατε όλοι Πέρας. Απορρίπτεται. 19-19. Καταπίπτει 48. 49 πάμε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά έλεγχος για την 52 ψήφισαν το όλοι πέρας ...17-20 απορρίπτωτα. Compromise 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται έλεγχος έλεγχος για την τροπολογία 3 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, έλεγχος για την τέσσερα. Πέρας. Δεκαοκτώ με δεκαεπτά εγκρίνεται. Πενήντα εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα χρησιμοποιώντας τις κάρτες, τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες, πέρας. «34 υπέρ, 4 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, παρακαλώ, θα ήθελα να καθίσετε για να συνεχίσουμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Σημείο 8 έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Για την προσωπία της Επιτροπής Λίμπε στην Ελλάδα από 28 με 31 Οκτωβρίου του 2012. Έχουμε σχέδιο εκθέσεως αντιπροσωπείας. Όπως ξέρετε συνάδελφοι έγινε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή στις 19 Ιουνίου. Ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός για την Προστασία του Πολίτη, ήταν εδώ και μετά από τη συζήτηση έχουμε την έκθεση της αντιπροσωπείας. Δυστυχώς ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας, ο κ. Μούλντερ, όπως ακούσαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Η κυρία Βέμπερ είχε την καλοσύνη να παρουσιάσει την έκθεση της αντιπροσωπείας η ε, κυρία Βίξτρομ. Κυρία Βέμπερ μου λέγανε, ξέρω εγώ. Συγγνώμη κυρία Βίξτρομ. Τέλο πάντων από W ξεκινάνε τα ονόματα. να Να τα βρείτε. Κυρία Βίξτρομ. Γιατί αυτή η περιπτώση μιλήστε πρώτη για την έκθεση αντιπροσωπείας και μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα Πρόεδρος. Είναι πάντα Ανανεωτικέ οι καινοτομίε ακόμα και σε μια επιτροπή σαν τη δική μα. Εκ μέρου του Γιάνν Μούλτερ παίρνω το λόγο με τα χαράς και εφόσον ο Γιάνν Μούλτερ προείδρευε της αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καλώς ορίζει αυτή την έκθεση διότι σωστά αντικατοπτρίζει τα όσα είδαν τα μέλη της αντιπροσωπείας στην αποστολή αυτή στην Ελλάδα. Ο κύριος Μούντερ θεωρεί ότι μπορεί εν γέννη να υποστηριχθεί η έκθεση και ευχαριστεί τα μέλη της αντιπροσωπείας για το θετικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερατε Πρόεδρε, συζητήθηκε το θέμα μέσω email Έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών που ήταν στην αντιπροσωπεία του Οκτωβρίου και πρότεινα και τροπολογίε που συμπεριλήφθησαν. Σαν επικεφαλή αντιπροσωπεία ΛΥΜΠΕ πρότεινε δύο αλλαγέ ο Γιάνν Μούλτερ. Πρώτα απ' όλα οι παραθέσει να διαγραφούν των, των όσων είπαν τα μέλη στην έκθεση για να παρουσιάζονται απλώ τα στοιχεία και αναφέρονται στο κείμενο οι θέσει των ομάδων για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Δεν ήμουν στην αντιπροσωπεία όμως μου αρέσει πολύ η Ελλάδα και έχω κάνει άλλες αποστολές στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι έγινε αυτή η αποστολή και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που πραγματοποίησαμε αυτή την αποστολή. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλεια. Σχόλια για την επίσκεψη, για τα αποτελέσματα που αναφέρονται. Ορίστε θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την έκθεση και την υπερψηφίζω, την υποστηρίζω. Ε, κυρία Γκίου, απλώς δεν συμμετείχα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ καλά οργανωμένη αυτή η αποστολή. Νομίζω τελικά αποτελέσματα είναι λεπτομερέστατα και λαμβάνουν υπόψη αυτά που έγιναν Αυτές τις μέρες συμμερίζουμε το συνέστημα του κυρίου Μούλτερ για τη διαγραφή κάποιων σχολείων όχι που δεν είχαν θέση αλλά ήταν αντιφατικά τα σχόλια. Και λαμβάνει υπόψη το κείμενο ακριβώς λεπτόμερος και υποστηρίζω λοιπόν αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο κ. παπα Και εγώ να προσθέσω ότι υποστηρίζουμε το κείμενο αυτό. Θα ήθελα δύο γενικά σχόλια να κάνω. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν εύκολο να σχολιάσουμε το κείμενο εμείς μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό δεν φταίει πάντα η διοίκηση. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Το συζητήσαμε και με τον Υπουργό αυτό. Αποτελεί πραγματικότητα. Πριν από δύο εβδομάδες το συζητήσαμε. Είναι απειρχιωμένα κάποια στοιχεία που παρατίθενται λόγω προσφάτων εξελίξεων. Ε, έχουμε κάποια σχόλια, ανταλλάσσουμε email όσον αφορά τα σχόλια για κάποια κέντρα κράτηση που έχουν κλείσει πια στην Ελλάδα. Μετά από σχόλια και τη δική μα αντιπροσωπεία. Πιθανότατα λοιπόν σε μελλοντικές αντιπροσωπείες θα είναι σημαντικό να προβλέπετε χρονοδιάγραμμα. Το συμφωνήσουμε και μεταξύ μας. Πότε θα ετοιμάζετε το τελικό κείμενο της έκθεσης. Για να ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να σχολιάσουμε το κείμενο. Να επαγρυπνούμε. Και να βλέπουμε και να εξετάζουμε κατά πόσο το κείμενο της εκθέσεως είναι αντικειμενικό. Δεύτερον, Καμιά φορά όλοι όσοι συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους αντιπροσωπείες για τη διαπίστωση γεγονότων και στοιχείων πρέπει να συμφωνούμε, και είναι σημαντικό αυτό, επί των κρισίμων σημείων που θέλουμε να υπογραμμίσουμε κάθε φορά. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, να λέμε θα δούμε το ένα μέρος, το άλλο μέρος, το παράλληλο. Ας πούμε ότι κάποιος έρχεται εδώ και βλέπει ότι λείπει ένα φως, σε ένα σπίτι λείπει ένας γλόμπος. Δεν σωστό να λέει έκθεση ότι λείπει ένα φως, ένας γλόμπο, ενώ υπάρχουν άλλοι 200 γλόμποι που λειτουργούν. Δημιουργείται ίσω λανθασμένη εικόνα για την πραγματικότητα έτσι. Άρα είναι σημαντικό να προσπαθούμε να συμφωνήσουμε επί κρισίμων σημείων. Και δεν το αναφέρω αυτό μόνο για αυτή την έκθεση. Και ευχαριστώ και τους συμβούλους μας για την συνεισφορά τους και το πώς αντιμετώπισαν τη σύνταξη της εκθέσεως. Δεν ήταν εύκολο για μας μετά από τόσο καιρό να βρούμε μια ισορροπία. Ευχαριστώ για την ισορροπία που βρήκαμε, τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μούλτερ. Υπήρξε σοφό στην προσέγγιση του, σοφά τα όσα πρότεινε. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της ε, αντιπροσωπείας και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να συνταχθεί σωστά αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση εμπεριέχει ορισμένα στοιχεία τα οποία ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι εγώ τώρα μόλις έλαβα την έκθεση και δεν πρόλαβα να την ε, διαβάσω. Αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο έχουν επιληθεί τα προβλήματα τα οποία ε, διότι η επίσκεψη έγινε εδώ και ένα χρόνο. Και θα ήταν ε, ε, ενδιαφέρον να δούμε τι επιλήθηκε, δηλαδή να αποτιμήσουμε και να δούμε κατά πόσο η συλλογιστική που μας διείπε τότε ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, διότι Υπάρχουν προβλήματα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά και κέντρα κράτησης σε άλλες χώρες. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε ποια μέτρα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο είναι ε, αποτελεσματικά, διότι στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο να προσδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή του μετανάστη. Άρα όλα αυτά τα πρόσωπα που ήταν σε κέντρα κράτησης ε, δεν είχαν δυνατότητα ταύτισης ή αναγνώρισης. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα αργή, αλλά αυτό δεν είναι θέμα της Ελλάδας, είναι διεθνές ζήτημα. Στα κέντρα αυτά κράτησης χρειάζεται πολύς χρόνος για την ταύτιση και την αναγνώριση. Και το αρχικό διάστημα των τριών μηνών παρατάθηκε στους έξι μήνες. Δηλαδή σε άλλες χώρες υπάρχουν άλλες προθεσμίες. Στη δική μας είναι των 24 ημερών. Αυτό που έχει σημασία είναι η αναγνώριση και η ταύτιση αυτών που βρίσκονται στα κέντρα. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση αναγνώρισης. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεψε ώστε να μειωθούν αυτές οι προθεσμίες. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο εντοπίσαμε ήταν η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων για τους ετούντες άσυλο. Είτε πρόκειται για παράνομους μετανάστες είτε όχι. Φαίνονται όμως ως ετούντες άσυλο καταρχήν. Και η Ελλάδα αποφάσισε να περάσει την αρμοδιότητα από τις αστυνομικές αρχές σε ένα ειδικό σώμα εμπειρογνωμόνων. Δέξαμε κατά πόσο έγινε αυτή η μετάβαση αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα. Κατά πόσο συστάθηκε δηλαδή αυτό το ειδικό σώμα για τους ετούντες άσυλο. Γι' αυτό αφορά και άλλες χώρες. Επίσης δεν υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής ε, ε, στην Τουρκία και δεν ε, χορηγούνται θεωρήσεις γιατί είναι δύσκολο να περάσουν, δεν μπορούν να περάσουν αυτοί οι μετανάστες χωρίς θεώρηση στην Τουρκία. Και βεβαίως και με την κατάσταση της Συρίας έχει οξυνθεί το θέμα της μετανάστευσης Ξέρουμε δηλαδή τώρα και ότι και η θαλάσσια μεταφορά χρησιμοποιείται περισσότερο και μετά. Ε, και κλείσανε δύο κέντρα μετά από την επίσκεψή μας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι εξαιτία μάλλον χάριν σε αυτή την ε, επίσκεψη επιλήθηκαν ορισμένα ζητήματα, κλείσαν δύο κέντρα, αλλά ως προς άλλα ζητήματα, ανοιχτά ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί και πόσο χρειάζεται ακόμα την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποιους τομείς. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου θα ήθελα να επανέλθει σε ορισμένα σημεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομέρα Λόπες ε, κοιτούσε μένα κατά τις δηλώσεις αυτές. Εγώ δεν εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση, μπορώ να σας δώσω όμως ορισμένε πληροφορίες. Στην εισαγωγή μου δεν ήθελα να μπω στην ουσία γιατί είδα ότι και άλλοι συνάδελφοι δεν το έκαναν. Αλλά εντάχει θα ήθελα να σας πω ότι πολλά από τα ζητήματα που έθιξε η κυρία Ρομέρο Λόπες απαντήθηκαν από τον Υπουργό δύο εβδομάδες πριν στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η έκθεση αυτή, μετά από τα σχόλια και τις διαπραγματεύσεις με τις πολιτικές ομάδες, δείχνει ότι έχουν επιτευχθεί θετικές εξελίξεις το τελευταίο χρόνο και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από τις ελληνικές αρχές να τηρούνται επαρκώς τα δικαιώματα όλων των ε, προσώπων από, τις τρίτες, από τρίτες χώρες και να καλύπτονται και οι ανάγκες τους. Βεβαίως δεν ισχύει αυτό πάντα όταν έχουμε μεγάλες ροές Υπάρχουν χάσματα, υπάρχουν κένα και θα ήθελα επίσης να πω ότι οι θετικές αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν οφείλονται στο γεγονός ότι ορισμένες αντιπροσωπείες ή εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν στην Ελλάδα για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα, μια εθνική στρατηγική και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εξέλιξεις και όταν ε, γίνονται επικρίσεις, αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία για τις ελληνικές αρχές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βεβαίως, υπάρχει και η νέα υπηρεσία χορήγησης ασύλου που έχει καταστεί λειτουργική mm. και ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις ε, θα μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Γι' αυτό ε, τόνισα ότι σε αυτή την έκθεση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάχρηση ασύλου από κατοίκους τρίτων χωρών προσπαθούν να βρουν συγκεκριμένα μονοπάτια όπως αυτοί που προωθούν το λαθρεμπόριο για παράδειγμα και χρησιμοποιούν αυτά τα μονοπάτια για να φτάσουν στους στόχους τους. Ε, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες του Νότου γενικότερα υπάρχουν θέματα στο εγγύς μέλλον προβλέπονται μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Ελπίζουμε μετά από αυτά τα σχόλια και τις αντιπροσωπείες στις χώρες που μεταβαίνουμε, Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα, την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούμε στην Ισπανία για τη Frontex. Ας ελπίσουμε ότι μετά από όλα αυτά τα σχόλια θα συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περισσότερες προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν για να υποστηρίξουμε εκείνους που το χρειάζονται. Να υπάρχει καλύτερος επιμερισμός ε, ε, καθηκόντων και να μην αποτελεί ευσεβή πόθο μόνο αυτός ο επιμερισμός, αλληλεγγύης, αυτός ο επιμερισμός αλληλεγγύης που δεν υπάρχει έμπρακτα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Η έκθεση θα εγκριθεί στα πρακτικά της επόμενης συνάντησης της ΛΥΜΠΕΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείο 9. Προτρέχουμε κάπως. Ο κύριος Δίας Δεμέρα κάθεται στη θέση του. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου 539 του 2001 σε σχέση με την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ε, από υπηκόους τρίτων χωρών. Ο κύριος Δίας Τεμέρα θα μας πει πώς έχει η έκβαση των διαπραγματεύσεων και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη που το επιθυμούν καθώς και στην Επιτροπή. Και βεβαίως και σε εκπροσώπους της ε, Προεδρίας αν το επιθυμούν. Ο κύριος Δίας Δεμέρα σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβω το λόγο μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης ε, διαφάνειας έτσι ώστε να σας δώσω πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης, δηλαδή πώς έχει η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Συμβουλίου 539 του 2001. Καταρχήν, μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων και οκτώ 8 τριμερείς διαλόγους, 8 των σκιουδών και 7 τεχνικές ε, συναντήσεις, 18 συναντήσεις με τους συνεργάτες και τους βοηθούς και πολλές συναντήσεις με τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αρχίσαμε υπό Ουγγρική Προεδρία, Πολωνική Κυπριακή και φτάσαμε και στην Ιρλανδική. Τον τριμερή διάλογο της 25ης Ιουνίου φτάσαμε σε μία συμφωνία με πλειοψηφία του Συμβουλίου με το ΕΛΚ, Φιλελευθέρους και τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Σε αυτή τη συμφωνία αναφερόμαστε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πάντες για την προσπάθεια που έχει καταβληθεί ιδιαίτερα από την Ιρλανδική Προεδρία που οδήγησε στην ομοφωνία του Συμβουλίου. Λοιπόν, το κείμενο λαμβάνει υπόψη την πλειοψηφία των σημείων που απέτησε το Κοινοβούλιο από την απαρχή των διαπραγματεύσεων. Το κείμενο αυτό αυτό είναι πανομοιότυπο με ορισμένες βελτιώσεις με βάση το συμβιβασμό του Δεκεμβρίου μεταξύ σοσιαλδημοκρατών, ΕΛΚ, φιλελευθέρων και Ευρωπαίων συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Άρα σας παρουσιάζω το ίδιο κείμενο του συμβιβασμού με ορισμένες βελτιώσεις θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εργασία όλων των σκιωδών. Ήταν μία συνεχής ακριβής εργασία και μας διείπε πνεύμα συμβιβασμού. Φτάσαμε λοιπόν σε συμβιβασμού στα εξή θέματα. Θεώρηση για τα μέλη διάσωσης για το προσωπικό ε, φροντιστές ε, αεροπλάνων, για τις θαλάσσιες μεταφορές και αυτά τα θέματα ίσως φαίνονται ίσονο σημασίας αλλά δεν είναι. Γιατί αναφερόμαστε στην ε, διαδικασία αμοιβαιότητας και αναστολής ως προς το θέμα της αμοιβαιότητας. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη επί του θέματος και θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα αποδοτικό και αλληλέγγυο μέσο το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις ε, εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια, τη στιγμή που ένα τρίτο κράτος ε, ζητά θεώρηση, η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να προβάλλει όλες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να επιλυθεί το ζήτημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προτείνει την προσωρινή αναστολή χορήγησης θεώρησης. Το σημείο κλειδί είναι ότι το θέμα είναι στη διακριτική ευχαίρεια της Επιτροπής. Δεν αποτελεί υποχρέωσή της. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Είναι διαφορετικό βεβαίως όταν παρέλθουν τα δύο χρόνια από τότε που ανακύπτει το πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο όρισε αυτό το διάστημα των δύο ετών έτσι ώστε να τεθεί εν λειτουργία μία αυτόματη αμοιβαιότητα, διαδικασία αμοιβαιότητας μέσα από μία νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με το Συμβούλιο. Στα δύο χρόνια λοιπόν η Επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να ζητήσει την αναστολή θεώρησης για ε, υπηκόους τρίτων χωρών ε, χρησιμοποιώντας μία κατεξιοδότηση πράξη. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα. Δηλαδή όχι μόνο χρησιμοποιούνται οι κατεξουσιοδότηση πράξεις αλλά φτάνουμε σε αυτή την αυτόματη απαλλαγή. Όταν αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις, κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο τώρα, χάρη στην εργασία που ε, προωθήσαμε από κοινού, αυτό αποτελεί πραγματικότητα. Θα ήθελα να μιλήσω και για το μηχανισμό αναστολής. Φτάσαμε σε σημαντικά ε, βήματα τα οποία δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο. Δηλαδή υπάρχουν ε, ρήτρες διασφάλισης την οποία θα, τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή κατά την ε, προσωρινή αναστολή χορήγησης θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπετε, πρόκειται για μία λεπτή ισορροπία. δύναμη αυτού του συμβιβασμού. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε δύο άλλα ζητήματα, τα οποία θα ήθελα να σας επεξηγήσω και να σας γνωστοποιήσω. Το πρώτο είναι το εξής. Το κείμενο προβλέπει να υπάρξει μία ρήτρα αναθεώρησης ε, μετά από 7 χρόνια. Από τότε που θα προβλεφθεί ε, απαλλαγή χορήγης θεώρησης. Και το επεξηγώ. Αυτή η προθεσμία είναι πολύ καλύτερη από την αρχικά προβλεπόμενη ένα χρόνο πριν ή αυτή που πρότειναν μερικοί άλλοι, δηλαδή τρία χρόνια. Και αυτό για ποιο λόγο. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα πιστικά. Δείχνουν ότι κατά τα δύο πρώτα έτη μετά από την ε, απελευθέρωση από το καθεστώς θεωρήσεων, τότε ορίζονται και αναγνωρίζονται θέματα μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γι' αυτό κατά την άποψη μου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής προθεσμία έτσι ώστε η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις τρίτων χωρών να συνεργαστούν για να επιληθεί αυτό το θέμα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ότι μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, τότε μειώνεται ο όγκος των μεταναστευτικών ορών. Αυτό είναι αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Και αν ρίξετε μια ματιά στις εκθέσεις για τα Βαλκάνια, το βλέπετε αυτό. Άρα χρειάζεται χρονικό διάστημα για τα κράτη μέλη ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχανισμό. Γι' αυτό, εάν προβλέπονταν μόνο τρία χρόνια, τα κράτη θα προέβλεπαν τον μηχανισμό αναστολής χωρίς να προστρέξουν στη διαπραγμάτευση ακριβώς επειδή θα ήταν πολύ μικρή η προθεσμία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ρήτρα για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των άλλων χωρών, τη στιγμή που υπάρχει αυτό το καθεστώς απελευθέρωσης. Και έτσι αυτός ο μηχανισμός θα είχε κατασταλτική ισχύ, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε με την προθεσμία των 7 ετών. Έτσι δεν υφίστανται πίεση ούτε τα κρατη ούτε οι τρίτες χώρες και έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τα κατάλληλα μέσα για την επίλυση του ζητήματος. Γιατί τα προβλήματα αυτά πάντα ανακύπτουν τη στιγμή που υπάρχει απελευθέρωση. Βλέπουμε ότι χρειάζεται έλεγχος στα σύνορα και αυτό για πάνω από πέντε χρόνια. Έτσι θα εξαλειφθούν τα προβλήματα της απελευθέρωσης από το καθεστώς αυτό. Βεβαίως θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την πολιτική θεωρήσεων, τη σωστή πολιτική αντιμετώπιση των θεωρήσεων. θα χρησιμοποιήσουμε και τις εκτελεστικές ε, πράξεις. Αλλά εξ αρχής το Κοινοβούλιο ήθελε ομόφωνα να χρησιμοποιηθούν εκτελεστικές ε, πράξεις όπως όρισαν οι τροπολογίες των ε, πολιτικών ομάδων και το αρχικό κείμενο του Απριλίου του 2012 της ΛΥΜΠΕ, καθώς και η συμφωνία μεταξύ σοσιαλδημοκρατών, ΕΛΚ, ε, Πρασίνων, Φιλελευθέρων και του, των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Όλοι θέλουμε λοιπόν εκτελεστικές πράξεις και ε, η Ιρλανδική Προεδρία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και δεν μπορεί να κοφεύει. Αυτή... Αυτό ήταν ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Εάν ε, συμπεριλάβουμε τις, ε, ε, συμπεριλάβαμε τις κατεξουσιοδότηση πράξη, αυτό το κάναμε για να έχουμε ένα μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να δούμε τι θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε. Άρα το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων ή εκτελεστικών πράξεων είναι ένα ε, θέμα οριζόντιας ερμηνείας το οποίο θα δούμε κατά περίπτωση. Δεν θέλω να χάνουμε το, τον ευρύτερο ορίζοντα, δηλαδή την πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Έτσι έχει η κατάσταση και ο εισηγητής λοιπόν θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόοδο έτσι ώστε να ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο στις 8 και 9 από όσο γνωρίζω. Μετά από συζήτηση βεβαίως. Έτσι ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας διαφάνειας και θα ήθελα να ακούσω την απόψη των συναδέλφων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία που με βοήθησε ιδιαίτερα και ιδιαίτερα του Σκιώδη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία τους. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Θα ζητήσω τώρα από τους σκιώδης εισηγητές που βρίσκονται εδώ να λάβουν το λόγο να σας αναφέρω όμως πρώτα ότι υπάρχουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Συμβουλίου για να μας απαντήσουν μετά τους συναδέλφους. Κύριε Φάιον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή Βρίσκομαι σε μια αρκετά λεπτή θέση αυτή τη στιγμή, διότι οι διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες των κανονισμών συνεχίζονται εδώ και δύο χρόνια τώρα και υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ε, ήμασταν πολύ κοντά σε συμφωνία και είχαμε εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Είχαμε μάλιστα καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία το Δεκέμβριο όμως ε, το θέμα εμποδίστηκε από το Συμβούλιο. Επίσης, ε, πολλές φορές ε, πέσαμε θύματα εκβιασμού, αν θυμάστε καλά, που αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και στο τελευταία στάδια των συνομιλιών θυμάμαι ότι ορισμένοι Αμερικανοί διπλωμάτες μας πίεσαν πάρα πολύ όσον αφορά τον μηχανισμό αμοιβαιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτή η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι προϊόν ομοφωνίας από τον τελευταίο τριμερή διάλογο και πιστεύω ότι αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι εξισορροπημένος συμβιβασμός, δεν είναι καλός συμβιβασμός, το αντίθετο μάλιστα. Και να σας πω καταρχάς ότι το πιο σημαντικό φυσικά είναι το θέμα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση όσον αφορά τις ερήτρες αναστολής. Τον Απρίλιο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ψηφίσαμε την δική μας ενισχυμένη θέση, η οποία υποστηρίχθηκε σχεδόν ομόφωνα το Μάρτιο από τους κοιόδης εισηγητές, ε, όπου προβλέπαμε πράξεις κατά εξουσιοδότηση και για τους δύο μηχανισμούς, και για τις ερήτρες αμοιβαιότητας και για τις ερήτρες αναστολής. Μετά από λίγο καιρό, όπως ακούσατε, προς έκπληξη της ομάδας μας, ο εισηγητής δέχτηκε ένα κείμενο του Συμβουλίου, το οποίο είναι αντίθετο στην θέση του ΕΛΚ και της Επιτροπής και της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία προβλέπει συναπόφαση. Με άλλα λόγια, δυστυχώς ο εισηγητής ε, άφησε το θέμα των πράξεων εξουσιοδότησης στον μηχανισμό αναστολής. Αυτό τι σημαίνει, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απανείται τις εξουσίες που του έχει δώσει η συνθήκη της Λισαβόνας και το Συμβούλιο αγνοεί απλά και καθαρά το Κοινοβούλιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, δυστυχώς φοβάμαι ότι τώρα διακυβεύονται πολλά από τα οποία, τα οποία συζητούμε τώρα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ποια θα είναι η συνέπεια εάν ψηφίσουμε τον Σεπτέμβριο σε σημερινές συμβίβας, τον σημερινό συμβιβασμό. Πολύ φοβάμαι ότι ο μηχανισμός αναστολής θα τεθεί σε λειτουργία για πάρα πολλές ε, χώρες και πολλές ε, φορές, σε πολλές περιπτώσεις θα επανεισαχθούν ε, οι θεωρήσεις σε πολλές χώρες. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα μας ήταν η χαλάρωση των κανόνων υποχρέωσης θεώρησης, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Και ας είμαστε ξεκάθαροι, 7 χρόνια επεξεργαζόμαστε αυτό το έγγραφο, 3 χρόνια βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις και γιατί θέλουν τα ορισμένα κράτη-μέλη να επαναφέρουν τις ε, θεωρήσεις ε, για ορισμένες χώρες Φυσικά, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ετούντων άσυλο στο μεταξύ, όμως τώρα αυτός ο αριθμός μειώνεται. Ωστόσο, επιμένουν οι, τα ρατσιστικά και εθνικιστικά σχόλια και δηλώσεις και αυτό πιστεύω τίνει να ε, καταχραστεί τις ε, εξουσίες και τις ε, αρμοδιότητές μας και να χαθεί η ευρωπαϊκή προοπτική από μπροστά μας. Επίσης, να πω στους συναδέλφους οι οποίοι πιστεύουν ότι βελτιώνουμε τον μηχανισμό αμοιβαιότητας να είστε βέβαιοι, βασισμένοι σε αυτόν τον συμβιβασμό και βασισμένοι στην επιστολή που έχουμε δει όλοι μας, η οποία διέρευσε. Η αμοιβαιότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ στην περίπτωση του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω εδώ, καταρχάς, αυτό που θεωρώ σημαντικό. Το θέμα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με πολλούς εφακέλους στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή. Πρέπει να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική θεωρήσεων ήταν πάντα κομμάτι των αρμοδιοντήτων μας και δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την ε, υπεράσπιση και άμυνα των Ευρωπαίων πολιτών για τα πιο θεμελιώδη και βασικά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να καταψηφίσουμε την πρόταση το Σεπτέμβριο στην πρώτη ανάγνωση και αυτό θα επιτρέψει και στα δύο θεσμικά όργανα να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να οδηγηθούν σε μια καλύτερη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βέιπα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή μας για αυτή την ε, συνεχή δουλειά και συνεχής προσπάθειες για αυτό το θέμα. Στην ε, αρχή ήμασταν ε, σε τελείως διαφορετική θέση από αυτή που έχουμε καταλήξει τώρα και ο εισηγητής μας έχει στηρίξει πάρα πολλές απόψεις όχι μόνο των σκιωδών εισηγητών αλλά και άλλων συναδέλφων οι οποίοι συνεργάστηκαν για αυτό το θέμα. Τώρα, επί της ουσίας και επί της διαδικασίας και όσο με το ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, θα ήθελα να σας πω μερικά σύντομα σχόλια. Πιστεύω πως με όλο το σεβασμό προς την Επιτροπή, ε, πιστεύω πως πολύ καλύτερα θα ήταν να είχαμε διαφορετικά τα πράγματα. Έχαμε μία ανακοίνωση για την αναστολή των θεωρήσεων και μία άλλη ανακοίνωση για την αμοιβαιότητα. Αυτή ήταν και η εφετηρία μας. Και μετά όλα αυτά τα δύο συγχωνεύτηκαν. Και επίσης, γεγονός είναι ότι και εγώ και ο συνάδελφος Άλεξ Άλβαρο και η Τάνια καταθέσαμε μία τροπολογία η οποία ήταν πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων και χωρίς την τροπολογία αυτή θα είχαμε ολοκληρώσει το θέμα, δεν ξέρω, ενδεχομένω και πριν από δύο χρόνια, διότι η αλήθεια είναι ότι μήνες επιμηνών συζητούσαμε την αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις. Και ευθύ εξ αρχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα δεν ζήτησε πράξεις κατά εξουσιοδότηση για την αναστολή εκτός θεωρήσεων. Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις συμφωνήσαμε μεταξύ μας για εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά την αναστολή των θεωρήσεων και τότε θεωρούταν ότι ό,τι έχουμε συμφωνήσει δεν θα το ξανανοίξουμε. Μετά η διάσκεψη των Προέδρων, έξι μήνες αργότερα, αποφάσισε για λόγους πολιτικής ότι θέλουμε πράξεις κατά εξουσιοδότηση γενικά. Όχι, δεν πιστεύω ότι χωρίς αυτές θα διακινδυνεύσει η θέση μας και οι αρμοδιότητές μας. Αυτή ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων και είχε πολιτικό χαρακτήρα και απόχρωση. Διότι η αλήθεια είναι ότι είτε με πράξεις κατά εξουσιοδότηση, είτε με εκτελεστικές πράξεις, η απόφαση αυτή δεν είναι πλέον στο χέρι των κρατών μελών, αλλά στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι που θέλαμε να διασφαλίσουμε, ότι δηλαδή στο μέλλον θα αποτρέψουμε και θα αποφύγουμε οποιαδήποτε πιθανότητα κατάχρησης από κάποιο κράτος μέλος που θέλει να επαναφέρει τις θεωρήσεις. Και Επίσης, πάλι με όλο τον σεβασμό για τους φίλους μας από τις βαλκανικές χώρες, η αλήθεια είναι ότι όταν εμείς νομοθετούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, νομοθετούμε γενικώ. Αυτό ε, είναι το θέμα του φακέλου αυτού. Δεν απευθύνεται ιδιαίτερα στους κατοίκους των Βαλκανικών χωρών, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουμε κατά νου ορισμένες από τις ε, εντός εισαγωγικών απειλές από κάποια κράτη-μέλη, έτσι όπως έχουν αναφερθεί. Στα πλαίσια της υφισταμένης συμφωνίας, όταν λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια απόφαση, ακόμα και αν είναι για 7 χρόνια, είναι αυτά τα 7 χρόνια κάτι που θα πρέπει να προκύψει μετά από εκτιμήσεις της Επιτροπής. Είναι εκτίμηση της Επιτροπής. Εάν εδώ υπερψηφίσουμε αυτό το φάκελο, στην ουσία τι θα γίνει. Κανένα κρατός μέλος δεν θα μπορεί να επαναφέρει ε, την υποχρέωση θεώρησης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να το κάνουν είναι αυτός εδώ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους ε, πολίτες των ε, δυτικών βαλκανικών χωρών εάν καταψηφίσουμε το φάκελο αυτό. Τώρα, κατόπιν τούτου να πω ότι η απόφαση πιστεύω πως και φοβάμαι μάλιστα πως θα είναι πάλι πολιτική και πως πάλι θα πάμε στην διάσκεψη των Προέδρων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παροτρύνω τώρα τους σοσιαλιστές να ξανασκεφτούν την προσέγγισή τους για την ουσία της συμφωνίας αυτής και να δουν ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλουν. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους κατοικούς των Βαλκανίων ή όχι. Εάν ναι, τότε δεν καταλαβαίνω πώς θα το κάνουμε αυτό χωρίς να, να αναλάβουμε δράση, να αφήσουμε την κατάσταση όπως έχει τώρα, όπου το κάθε κράτος μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπερψηφίσουμε λοιπόν. Αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις, τώρα ναι, έχουμε έναν ε, διπλό μηχανισμό και εκτελεστικές και πράξεις κατά εξουσιοδότηση, και εντάξει, ίσως ε, δεν ε, μας πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά όπως και να έχει μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ότι δεν συμφωνεί θα εκδοθεί. Δεν είναι η αμοιβαιότητα αυτό που θέλουμε, αλλά το, αυτό πιστεύω πως το μόνο που δείχνει είναι την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσποιείται και παριστάνει έναν σημαντικό παράγοντα, αλλά απέχει παρασάκας από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ντονόκ. Yes. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας, όπως ξέρετε, καταψήφισε Suspension. του μηχανισμού αναστολής. Αυτή είναι η βασική μας θέση. Ήμασταν επικοδομητικοί, προτείναμε κάποιες τροπολογίες όμως τη στιγμή αυτή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια συμφωνία τέτοια για το μηχανισμό αναστολής. Όσον αφορά την αμοιβαιότητα, έχει επιτευχθεί πρόοδος, καλή. Βασική μας ανησυχία είναι ο μηχανισμός αναστολής δεν θέλουμε αναστολή αυτή καθεαυτή και σίγουρα όχι μέσω κατοξισοδότηση, μέσω εφαρμοστικής πράξης μάλλον. Αυτή λοιπόν η θέση των σοσιαλιστών που τη γνωρίζει και ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Έντσου, θέλετε να μιλήσετε, το ξέρω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμέρα για αυτή την εξαιρετική του εργασία, για, το, για τα όσα κατάφερε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση των πολιτών μιας χώρας όπου δεν υπάρχει αμοιβαιότητα σχέσεων με, τα, με Καναδά και ΙΠΑ αυτούς τους πολίτες πρόσωπο. Νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη αυτή την ανώμαλη κατάσταση, ορισμένες τρίτες χώρες ε, δεν αναγνωρίζουν τα ίδια ε, δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη κατά περίπτωση για το καθοστός των ε, θεωρήσεων. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν ε, κατασταλτικοί μηχανισμοί ή δεσμευτικοί μηχανισμοί έναντι τρίτων χωρών, τότε δεν μπορεί να αντιδράσει ενωτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη επίσης δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα για την ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Δεν είχε βεβαίως και την κατάλληλη νομική βάση θεωρώ ότι αυτή η νέα ρήτρα αμοιβαιότητας μπορεί να αποκαταστήσει τα πράγματα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αξιοπρεπής και αποφασιστική με τους διεθνούς, διεθνείς εταίρους. Θεωρώ ότι η ρήτρα αμοιβαιότητας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός έτσι ώστε να υπάρχει η ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό ανεξάρτητα από τα πολιτικά ε, κόμματα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία με το σύμβολο. Ευχαριστώ. Κυρία Φαϊόν, θέλετε να επανέλθετε να σχολιάσω στα τα όσα είπε η Ρενάτε, συνάδελφος. Αφορά το ζήτημα της πολιτικής θεωρήσεων. Έχει ρυθμιστεί μέσω διαδικασία συναπόφαση διαδικασία θεωρήσεων και αν μέσω ρήτρα αναστολής παρατηθούμε από τις κατεξουσιοδότης συμπράξεις, αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα ρωτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί όταν θα ληφθεί απόφαση για επανεισαγωγή θεωρήσεων. Γι' αυτό το κίνδυνο μιλάω σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση που έχουμε διάφορες κυβερνήσεις που έχουν πλειοψηφία στο Συμβούλιο και θέλουν μέσω πλειοψηφίας να επαναφέρουν τις θεωρήσεις και όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια και για τους κανόνες έγκαινα έχουμε προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων. Σήμερα είναι διαδικασία συναπόφαση. Φοβούμαι ότι αν υπαναχωρήσουμε θα χάσουμε πολλά όσον αφορά το μελλοντικό προσανατολισμό που θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία θα πάρουν το λόγο και μετά θα ζητήσουμε το λόγο ξανά στον κύριο Διασδεημέρο στο τέλος για τυχόν σχόλια. Ο κύριος Παύλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συγητή, τον κύριο Ντίας Δημέρα, όπως και οι συνάδελφοί του για τη δουλειά που έκανε. Μακρές και δύσκολες ήταν οι διαπραγματεύσεις. Καλωσορίζουμε τη συμφωνία που φαίνεται ότι επετέφθη. Όμως η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το θέμα είναι πασίγνωστη. Πάντα θέλαμε να έχουμε εύρυθμο μηχανισμό για αμοιβαιότητα και αναστολή, αλλά οι δύο μηχανισμοί έπρεπε να είναι θεσμικά σωστοί και νομικά σωστοί. Και φοβούμε ότι αυτή η συμφωνία που βλέπουμε μας δημιουργεί προβλήματα, ακόμα προβλήματα. Κυρίως οι προβλεπόμενες εξουσιοδότηση συμπράξεις για τη δεύτερη φάση του μηχανισμού αμοιβαιότητας που προβλέπεται υποχρέωση που υπέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αθετήσει πράξη κατά εξουσιοδότηση, αυτό κατά την άποψή μα δεν ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπώς επιφυλάσσεται στον αφορά τη θέση τη. Εν ευθέτω χρόνο θα προβεί σε δήλωση επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της και των νομικών της μέσων. Παρ' όλα αυτά, να τονίσω εκ νέου ότι αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, γρήγορα. Έχει πολύ κρατήσει όλη η ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς δεν μπορεί να δεχτεί όμως ε, προτάσεις ή μηχανισμούς οι οποίοι δεν είναι νομικώς ορθοί. Δυστυχώς εκφράζουμε επιφύλαξη όσον αφορά τη θέση μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Προεδρία του Συμβουλίου ο κ. Στριουψατ έχει το λόγο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τις απόψεις της Προεδρίας. Χαιρόμαστε που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και κατεπήγον. Η Προεδρία θέλει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερο τον εισηγητή κ. Ντεμέρο και τους βοηθούς του και όλους όσους συμμετείχαν στην αποπεράτωση αυτής της συμφωνίας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και σας και ευχαριστούμε την Πολωνική, τη Δανέζικη και την Κυπριακή Προεδρία και πάνω απ' όλα την Ιρλανδική Προεδρία για τις καταβληθήσεις προσπάθειες. Την προσπάθεια που κατεβλήθηκε για καλό συμβιβασμό μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Τέλος, διαβεβαιώνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ότι η Προεδρία είναι έτοιμη πάντα να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως προανέφερα, αν ο κ. Δίας Δεμέιρο θέλει να πάρει το λόγο, είναι ευπρόσδεκτος. Ε, θα ήθελα μόνο για λόγους ευπρέπειας και ευγένειας να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα, διότι ο φάκελος αυτός μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό με αντιγνωμίες και ε, διάφορες ε, διαφωνίες γενικότερα. Επί της ουσίας θα πρέπει να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε μετά από συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι πριν από την ψηφοφορία να γίνει συζήτηση για να ακουστούν όλες οι απόψεις και να κριθούν από την Ολομέλεια. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ και να προβάλλω απόψεις ε, αν λάβουμε ε, ε, υπόψη και την εξέλιξη των συζητήσεων. Δεν θα ήθελα να προδικάσω την έκβαση και να ε, προδικάσω την έκβαση του άλλου στήματος ε, ως προς ε, μία θετική εξέλιξη. Αυτό που είναι εξαιρετικό πολλές φορές μπορεί να μετατραπεί στο ακριβώς αντίθετό του. Γι' αυτό πιστεύω ότι πολλές φορές ε, τα μαθηματικά μπορούν να μας δώσουν μία κάλυψη η οποία ε, δεν είναι πάντα επαρκής. Θα ήθελα να πω ότι καλύπτουμε όλες τις προσδοκίες ε, συμπεριλαμβάνοντας αυτά που προτείνει η Τάνια. Καλύπτονται από την απόφαση αυτή δηλαδή να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, διότι ξέρουμε πολύ καλά ρυθμιστικά πώς θα λειτουργήσει η πρόταση. Η πρόταση μπορεί να ψηφιστεί και να εγκριθεί. Μπορεί να απορριφθεί επίσης. Εάν γίνει το πρώτο, τότε θα φτάσουμε σε συμφωνία. Tendremos que ir a segunda Εάν όχι θα φτάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Μπας περιπτώσει όλες οι προσδοκίες καλύπτονται και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε, να συζητάμε και να συζητήσουμε εν ολομελία έτσι ώστε η συμφωνία αυτή στον τελευταίο τριμερί μεταξύ ΕΛΚ, Φιλελευθέρων και Βρετανών συντηρητικών να μπορέσει να εγκριθεί. Τώρα, ως προς θέση της Κομισιόν και του Συμβουλίου, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Επιτροπή θα κάνει μία δήλωση. Ο κύριος Ντεκάστερ μας ε, προείπε ότι αυτό ακριβώς θα κάνει. Η Προεδρία του Συμβουλίου, καταρχήν η Επιτροπή είπε ότι επιφυλάσσεται. Το ξέρουμε, δεν είναι κάτι το καινούριο. Ξέρουμε ότι θα γίνει μια δήλωση. Εάν όμως προχωρήσει αυτή η συμφωνία με επαρκή πλειοψηφία, θα είμαστε σε θέση να αγγιθούμε αυτό το σύστημα χορήγησης ασύλου και να ε, προστατεύσουμε και τα δύο μέρη, και τους Ευρωπαίους ε, πολίτες και τους ετούντες άσυλο. Και δεν νομίζω ότι, ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο το, την οποιαδήποτε πλευρά και δεν θα επανισαχθούν οι θεωρήσεις. Και αυτό το λέω με μεγάλη πεποίθηση. Ευχαριστώ τη Ρενάτε, την εκπρόσωπο των φιλελευθέρων για τα καλά της λόγια και πιστεύω ειλικρινά ότι ε, γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση και κατανοεί ότι το θέμα του διαδικού αυτού μηχανισμού στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και ισχύει Ρενάτε αυτό που είπες η διάσκεψη των Προέδρων δεν ερμηνεύει την νομιμότητα. Πρόκειται για μία διάφρωση, για μία δομή που οδηγεί σε μία ε, πολιτική γνωμοδότηση. Όμως ε, δεν ορίζει, δεν, είναι μία ε, δογματική αρχή. Εγώ τάσομαι υπέρ της συναπόφασης και των εξουσιών που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας και η κατεξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να κριθούν κατά περίπτωση, αντίθεση με αυτό που λέει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλές φορές πρέπει να χρησιμοποιηθούν η κατεξουσιοδότηση πράξης και ξέρετε πόσες φορές είμαι υπέρμαχος αυτών. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αρχή του το μη χείρων βέλτιστον. Γνωρίζω πολύ καλά τη θέση της κυρίας Ιαρόκα και της ε, πολιτικής της ε, ομάδας και του κυρίου Έντσου τη θέση γνωρίζω που εκπροσωπεί τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας ναι. λόγια και για τα σχόλιά σας. Μιλήσατε για έναν δεσμευτικό μηχανισμό, για ένα κατασταλτικό μηχανισμό ως προς τις ε, τρίτες ε, χώρες. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επισούρουμε την προσοχή και σε αυτό το, το θέμα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για τη συζήτηση αυτή και θα το ξαναδούμε το θέμα το Σεπτέμβριο. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντίας Δεμέρα για διαδικαστικό και τυπικό. Αν υποστηρίζει το αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβληθεί στην Ολομέλεια και η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα και το Συμβούλιο, αν επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα των θα στείλει μια επιστολή την τυπική που στέλνει στη Συμφωνία Πρώτη Ανάγνωση. Και σωστά είπατε ότι η έκθεση προβλέπεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Τελειώσαμε αυτή τη συνεδρία επιτροπής. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.